στο δικό μου τμήμα του έργου, τους χάρη, σχετικά ε, με τον ΦΠΑ, τον ενεργειακό φόρο, τον, την φορολόγηση των εταιριών ε, και την ενίσχυση την τελωνιακή για τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας και για την ασφάλεια ε, των προϊόντων. Είμαι εδώ για να παρουσιάσω ορισμένες πρωτοβουλίες σχετικά με τα τελωνία. Τον Μάρτιο με χαρά ακούσα τον κύριο Μάλκομ Χάρμπορ ότι η Επιτροπή αυτή αποφάσισε να δώσει υψηλό πολιτικό προφίλ στα τελωνία με μια έκθεση ιδίας πρωτοβουλίας για τον εξυγχρονισμό των τελωνίων. Νομίζω ο κύριος Σαλβίνη θα ασχοληθεί και είχατε χτες μια σύντομη ανταλλαγή απόψεως. Νομίζω ότι διαμέσου των τελωνίων μπορούμε να έχουμε μια καλή λειτουργία της Τελωνιακής Ένωσης που βρίσκεται στο επίκεντρο της εσωτερικής αγοράς. Έχουμε δύο βασικούς στόχους, να διευκολύνουμε την ροή των αγαθών για τους νόμιμους εμπόρες, ενώ ταυτόχρονα θα προστατεύουμε τους πολίτες έναντι οποιοδήποτε κινδύνου για την ασφάλειά τους. Θα πρέπει να αντιδρούν τα τελωνία αρκετά γρήγορα για να προλάβουν την ε, μεταφορά επικινδύνων ε, προϊόντων ε, που θέλουν να μπουν, να εισέλθουν στο έδαφος της Ευρωπαϊκής Ένωσης χωρίς να μπλοκάρουν την ροή των ασφαλών προϊόντων. Το είδαμε αυτό πρόσφατα το πόσο σημαντικό είναι με την πυρηνική κρίση στην Ιαπωνία. Θα πρέπει λοιπόν να υπάρξει στενή συνεργασία με τις αρχές ασφαλείας. Οι μου έλαβαν ορισμένες πρωτοβουλίες για να υποστηριχθούν οι τελωνιακές διοικησει των κρατών μελών, ούτως ώστε να ενισχυθούν τα μέτρα κατά των μολυσμένων προϊόντων από την Ιαπωνία. Πρώτον, παρέχουν καθοδήγηση στις εθνικές τελωνιακές ε, διοικήσεις για να προστατευθούν οι πολίτες. Δεύτερον, εξασφαλίζουν την καλή διάδοση των πληροφοριών για επικίνδυνα προϊόντα σε όλα, τα τελωνιακά γραφεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Μέχρι τώρα είχαμε πολύ ελαφριά επιφανειακή μόλυνση ενός περιορισμένου αριθμού εμπορευματοκιβωτίων. Ωστόσο, το feedback και τα αποτελέσματα απέδειξαν την υψηλή ικανότητα των τελωνίων της Ευρωπαϊκής Ένωσης για ταχύτατο συντονισμό τους ώστε να ενισχυθεί η συνοριακή προστασία εναντίον οποιοδήποτε επικινδύνου ε, φορτίου. Θα πρέπει λοιπόν όπως ε, να ακούσετε την έκκληση της Επιτροπής ε, για ε, πιο ενεργό ρόλο στο συντονισμό των δραστηριοτήτων παρακολούθησης εσωτερικών εθνικών αγορών και τελωνιακών αρχών. Το νομικό πλαίσιο υπάρχει και μπορούν, να μπορεί να δοθεί καθοδήγηση στις δικήσεις. Ακούστε τις προτάσεις για φέτος σχετικά με την νομοθετική ατζέντα των τελωνίων. Εχθές η Επιτροπή υιοθέτησε μια πρόταση για ένα νέο κανονισμό για την ενίσχυση την τελωνιακή των δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας. Είναι μέρος της νέας στρατηγικής της Ευρώπης στον τομέα αυτό και νομίζω ότι η Επιτροπή σας θα έχει ενεργό ρόλο στην παρακολούθηση αυτή του θέματος. Η πρόταση η τελωνιακή ανταποκρίνεται σε πρόσκληση του Συμβουλίου σχετικά με τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας. Η πρόταση αυτή εξυπηρετεί ε, σημαντικότερους στόχους, ε, κυρίως την ενίσχυση των δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας από τα τελωνία, ενώ θα προστατεύονται τα συμφέροντα των νομίμων ε, των θεμητών εμπόρων. Επιπλέον η ε, πρόταση αυτή απαντά στις ανησυχίες ε, που έχουν αναφερθεί σχετικά με τις μικρές αποστολές αγαθών που αποστέλλονται ταχυδρομικά και ε, παραβιάζουν τα, τις οδηγίες που υπάρχουν σχετικά με τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας. Επίσης έχουμε διαφορές με την Ινδία, την Βραζιλία, σχετικά με τα γενώσιμα τα οποία περνούν από την Ευρωπαϊκή Ένωση ενώ αφήνεται ανοιχτή η πόρτα για τις απομιμήσεις. Ελπίζουμε ότι η πρόταση αυτή θα υιοθετηθεί το 2012 ως φοροτιμή στην ενία αγορά. Οι δύο άλλες νομοθετικές προτεραιότητες για φέτος συνδέονται με τον εξυγχρονισμό των τελωνίων. Πρώτον, θα ασχοληθώ με τον εξυγχρονισμένο ε, τελωνιακό κώδικα και τις διατάξεις εφαρμογή του. Όπως ξέρετε, η Επιτροπή και οι τελωνιακές αρχές εργάζονται συνεχώς, ούτως ώστε τα τελωνία της Ευρωπαϊκής Ένωσης να εργάζονται ταχύτερα και καλύτερα. Η εξυγχρονισμός των διαδικασιών είναι βασική προτεραιότητα για να απαντήσουμε στις προκλήσεις της ευξημένης ανάγκης για ασφάλεια σε μια απελευθερωμένη παγκόσμια αγορά. Οι υπηρεσίες μου έχουν κάνει τον απολογισμό ε, των προεργασιών και έχουν ε, προσδιορίσει την εικόνα για την κοινή εφαρμογή του εξυγχρονισμένου τελωνιακού κώδικα από την Κομισιόν, από τα εθνικά τελωνία, από τις δικήσεις και τους εμπόρους. Λόγω όμως της οικονομικής ε, κρίσης Νομίζω ότι τα συστήματα δεν θα είναι έτοιμα πριν από τον Ιούνιο του 2013. Αξιολογώντας ε, την κατάσταση υπηρεσίας μου, ε, συμβουλεύτηκαν πάρα πολλά εμπλεκόμενα ε, μέρη, της εθνικές τελωνιακές Διοίκησης, τους εμπόρους και επίσης αυτήν την Επιτροπή. Μπορώ να επιβεβαιώσω σήμερα ότι θα προτείνω μια πρόταση στο τέλος του έτους. Οι τροπολογίες έχουν ε, τρεις στόχους. Ε, πρώτον, την αναβολή της ημερομηνίας εφαρμογής του κώδικα, ούτως ώστε να υπάρξει ρεαλιστική εφαρμογή των νέων ηλεκτρονικών διαδικασιών, ούτως ώστε τα βασικά ωφέλη που αναμένουμε από τον εξυγχρονισμό να υλοποιηθούν. Δεύτερον, να εναρμονιστεί ο κώδικας με τις διατάξεις της συνθήκης της Λισαβόνας. Αυτή η εναρμόνιση απαιτείται κυρίως σε σχέση με την ε, χρήση ε, των κατεξουσιοδότηση πράξεων ή των ε, πράξεων εφαρμογής της Κομισιόν. Και τρίτον, η διόρθωση ενός περιορισμένου αριθμού διατάξεων του κώδικα ε, που έχουν σχέση με στοιχεία που δεν ισχύουν πλέον λόγω των αλλαγών που εισήχθηκαν το 2008 στην νομοθεσία της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή που σχετίζονται με στοιχεία που είναι δύσκολο ή αδύνατο να εφαρμοστούν. Βεβαίως η άσκηση αυτή είναι δύσκολη και έχουμε την προθεσμία της 24ης Ιουνίου 2013. Η επιτυχία εξαρτάται από την κοινή κατανόηση μεταξύ των εμπλεκομένων μερών. Δεν, δεν, έχει, δεν έχει ιδιαίτερη σημασία να ξαναρχίσει η συζήτηση ε, για τον στόχο και για τις αρχές του εξυγχρονισμού της τελωνιακής νομοθεσίας και να επαναλάβουμε τις συζητήσεις μεταξύ 2005 και 2008. Θα είναι χάσιμο χρόνο και δεν πρέπει να ξεκάνουμε αυτό το οποίο έχει ήδη γίνει. Θα πρότεινα μια παρέμβαση περιορισμένη και στοχοθετημένη στον κώδικα και ε, συνεχής προσπάθειες για να οριστικοποιηθεί το σχέδιο ε, εφαρμοστικής νομοθεσίας το συντομότερο δυνατόν. Υπάρχει μεγάλη ευκαιρία εναρμόνισης των προσπαθειών μας ήδη τώρα, εφόσον η, δική σας ε, η έκθεση ιδίας πρωτοβουλίας για τον εξυγχρονισμό των τελωνίων μπορεί να αναπτύξει και να προσδιορίσει μια κοινή κατανόηση των στόχων και της εμβέλειας της άσκησης. Πάνω σε αυτή τη βάση, η Κομισιόν, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το Συμβούλιο και τα Εθνικά Τελωνία θα μπορέσουν να υλοποιήσουν ε, το κεφάλαιο για τον εξυγχρονισμό ε, της Τελωνιακής Ένωσης. Θα ήθελα τώρα να στραφώ στην τρίτη μου ε, προτεραιότητα σχετικά με τον διάδοχο του προγράμματος Τελωνία 2013. Τα προγράμματα αυτά βοηθούν τις ε, εθνικές τελωνιακές αρχές να συνδεθούν με συστήματα πληροφορικής και να βελτιώσουν τον τρόπο ανταλλαγής των πληροφοριών. Είναι στοιχεία που έχουν μεγάλη προστιθέμενη αξία στο πρόγραμμα, κυρίως όσον αφορά τα διευρωπαϊκά ε, δίκτυα τεχνολογίας που αντιπροσωπεύουν 75-80% του προπολογισμού. Οι πρόσφατες αξιολογήσεις έδειξαν ότι το αντίκτυπο του προγράμματος ε, ξεπερνάει το σχετικά μικρό προϋπολογισμό που έχει επενδυθεί σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Μίλησα την περασμένη εβδομάδα σε ένα φόρουμ γενικών διευθυντών τελωνίων και συζητήσαμε σχετικά με τις ε, προκλήσεις και συζητήσαμε πώς θα μπορούσαμε να έχουμε οικονομίες κλίμακας, περισσότερη προστιθέμενη αξία και πρέπει να εξετάσουμε πώς μπορούμε να εξασφαλίσουμε την διαθεσιμότητα του καταλήλου εξοπλισμού και υποδομών σε όλα τα κράτη-μέλη. Αυτό θα βοηθούσε να μοιραστούμε ε, τον φόρτο της εργασίας για την προστασία των εξωτερικών συνόρων που για γεωγραφικούς και ιστορικούς λόγους ε, είναι ε, βαρύτερο το φορτίο από ότι σε ορισμένα κράτη-μέλη από ό,τι σε άλλα. Η Επιτροπή ε, οριστικοποιεί την πρόταση για το επόμενο πλαίσιο ε, το χρηματοοικονομικό, το πολυετές, για να δούμε ποιοι είναι οι περιορισμοί για μελλοντικές πρωτοβουλίες. Εν τω μεταξύ, οι υπηρεσίες μου αξιολογούν τις επιπτώσεις όλων των επιλογών που έχουμε για το μελλοντικό πρόγραμμα των τελωνιών. Μπορούμε να περιμένουμε την πρόταση το τέλος του έτους, πιθανότερα τον Νοέμβριο. Κυρίες και κύριοι αξιότιμα μέλη, σας παρουσίασα μια γενική εικόνα των νομοθετικών προτάσεων που έχω ή θα παρουσιάσω κατά τη διάρκεια του έτους. Όλες αυτές οι προτάσεις ε, εμπνέονται από τις, ε, τα, τους διτούς στόχους διευκόλυνσης του νόμιμου εμπορίου και προστασίας των πολιτών για την ασφάλειά τους. Ελπίζω να συμμερίζεστε τους στόχους αυτούς και περιμένω ότι θα έχουμε μια καρποφόρα ανταλλαγή απόψεων. Σας ευχαριστώ για την προσοχή σας. Σας ευχαριστούμε και εμείς. Ε, είμαι σίγουρος ότι θα υπάρχουν ερωτήσεις. Οι συνάδελφοι άκουσαν με μεγάλη ενδιαφέρον αυτά που είχατε να πει. Αυτό που είναι σαφές είναι ότι είναι πάρα πολύ έγκαιρη η παρουσία σας, γιατί έχουμε και την ε, έκθεση του συναδέλφου που προβλέπεται για την πρώτη ανάγνωση. Και όλα αυτά εντάσσονται και στρατηγική του 2013. Έχω ένα σκιώδη ε, συγητή, την κυρία Ράπτη, που θέλει να υποβάλει μια ερώτηση. Σαλντεμόζου είναι γενικά για την ασφάλεια στον τομέα αυτό. Δύο ανθρώπου που γνωρίζουν πάρα πολύ καλά τα θέματα. Λοιπόν, θα συμβάλλουν ερωτήσει και όποιο άλλο θέλει να υποβάλει ερωτήσει, παρακαλώ να μα κάνει ένα συνέλο. Εμεί συσχίζουμε με την κυρία Ράπτη. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Το, το παίρνω το θέμα πάλι από την αρχή. Ε, ε βέβαια, ε, η εισήγηση του κυρίου Σεμέτα ε, μου δημιούργησε ευχάριστα συναισθήματα. Ε, την άκουσα πολύ ρεαλιστική και αυτό μου άρεσε. Ε, μου δημιούργησε όμως ταυτοχρόνως και ερωτήματα. Ε, το πρώτο ερώτημα που έχω είναι το εξής. Όλα αυτά πάρα πολύ καλά από την πλευρά της Κομισιόν. Επειδή όπως ξέρουμε εκτός από την Κομισιόν υπάρχει και το Συμβούλιο, ε, τι προβλέπουμε να γίνει με το Συμβούλιο. Έχουμε κάποια αίσθηση, κάποια μυρωδιά. Δηλαδή, ε, στα ζητήματα που θέτει ο ίδιος και τα οποία εμένα μου φαίνονται πάρα πολύ ρεαλιστικά, ε, έχω την αίσθηση ότι έχουμε ανάγκη τη στήριξη του Συμβουλίου. Δεν ξέρω, υπάρχει. Ε, και από εκεί και πέρα θα ήθελα, αν είναι δυνατόν βεβαίως, κάποιες περισσότερες λεπτομέρειες τόσο σε σχέση με τη χρονική αναβολή, όσο και σε σχέση με τον ε, κώδικα. Και ευχαριστώ πάρα πολύ. Μία-μία ίσως τις ερωτήσεις να τις πάρουμε και θα προσπαθήσω να απαντήσετε στην κυρία Ράπτη πρώτα. Ναι, ναι, θα προσπαθήσω να είμαι σύντομος. προτού να προτείνουμε την αναβολή της ισχύω του ε, συγχρόνου κώδικα για τα τελωνία, ήρθαμε σε επαφή με τις εθνικές αρχές, με τους εμπόρους, με τους άμεσα διαφερόμενους και αυτή η προσέγγιση που σας περιέγραψα κιόλα. έτυχε της ε, ομόβουνης θα έλεγα υποστήριξης όλων των ενδιαφερομένων στη διαδικασία αυτή και ελπίζω ότι θα μπορούμε να έχουμε στο Συμβούλιο επικοδομητική συνεργασία για το θέμα. Βέβαια υπάρχει πάντα ο κίνδυνος να ξανανοίξουν πολλές από τις ζητήσεις για τα επιμέρους θέματα του κώδικα. Και γι' αυτό εγώ θα ήθελα να προτείνω να περιοριστούν οι τροπολογίες αυτές του κώδικα στο ελάχιστο που είναι απολύτως απαραίτητο. Και αν τηρήσουμε αυτή την προσέγγιση, νομίζω ότι η διαδικασία στο Συμβούλιο θα μπορούσε πραγματικά να είναι λιγότερο δύσκολη από ό,τι μπορούσε να είναι, αν το πω έτσι. Χρονοδιάγραμμα. Ομολογώ ότι η εργασία για τους κώδικες και τις ε, εκτελεστικές διατάξεις δεν έχει σταματήσει και εργαζόμαστε σκληρά πάνω σε όλα τα θέματα που αφορούν την εφαρμογή του εξοργανισμού αυτού του ελληνικού κώδικα. Και η ιδέα είναι να έχουμε όλα τα απαραίτητα νομοθετικά έγγραφα και μέσα έτοιμα μέχρι τις 24 Ιουνίου 2017 για να έχουμε μόνο το θέμα της εφαρμογής από εκεί και πέρα. Είναι πολύ σημαντικό να λάβουμε υπόψη ότι οι εξελίξεις για το της ηλεκτρονικής του, του, του, IT τέλο πάντων, της πληροφορικής ε, θα πρέπει να έχουν ένα πολύ αυστηρό πλαίσιο για να μπορέσουμε να, να εργαστούμε στην εφαρμογή τους. Ίσως να μπορούμε να υποβάλουμε κάποιες συμπληρωματικές μετά ερωτήσεις. Η κυρία Σάλτερ Μόζερ όμως έχει χρόνο πρώτα. Σας ευχαριστώ πολύ Πρόεδρε. Και θα να ευχαριστώ και τον Επίτροπο για την πολύ καλή παρουσίαση του τομέα και για τα προβλεπόμενα μέτρα. Πολλοί πιστεύουν ότι το λιονίο είναι ένα βαρυτό τομέα, αλλά είναι πάρα πολύ σημαντικό για την εσωτερική αγορά να λειτουργεί καλά το τολωνίο. Αν θέλουμε μια καλή εσωτερική αγορά και ασφαλή προϊόντα, χρειαζόμαστε και καλά τελωνία και καλή συνεργασία στον τομέα. Και γι' αυτό χαίρομαι ιδιαίτερα που σας άκουσα να λέτε ότι η συνεργασία αφενός με τις θέσεις ε, ελέγχου, με τις υπηρεσίες ελέγχου της αγοράς, και αφετέρου με το τελωνίο προωθείται από τις δικές σας υπηρεσίες. Εγώ θέλω να ξέρω τώρα τι μορφή θα έχει αυτή η συνεργασία, τι έχετε ξεκινήσει. Ένα αυτό. Και δεύτερον, τι γίνεται με τους σπόρους για τα τελωνία. Όσον αφορά το τομέα της ε, επιτήρησης αγοράς, ξέρουμε ότι σε περίοδους κρίσης πολλά κρατημέλη έκαναν περικοπές αυτών των πόρων. Τα τελωνία τι έγινε. Είδα και εκεί περικοπέ των πόρων. Και αν ναι, τι κάνει η Κομισιόν για να εξασφαλίσει να μην έχουμε περισσότερα επικίνδυνα προϊόντα στην εσωτερική αγορά. Συμφωνώ απόλυτα. Ότι η Ταλωνία δίνουν την εντύπωση είναι πάρα πολύ τεχνικό θέμα. Βέβαια καταλαβαίνουμε πώς λειτουργούν τα τελωνία μόνο όταν παρουσιαστούν προβλήματα. Όσο τα πράγματα πηγαίνουν καλά, εκατομμύρια διαδικασιών χωρίς πρόβλημα, δεν καταλαβαίνει κανένας τι σημαίνει τελωνία. Και βέβαια είναι πάρα πολύ σημαντικά για το μέλλον της ιστορικής αγοράς. Το θέμα της ασφάλειας είναι πάρα πολύ κέριο. Και γι' αυτό έχουμε την απαραίτητη νομοθεσία και εργάζονται πάνω σε αυτό τα τελωνία. Τελειοποιούμε αυτή τη στιγμή κατευθυντήριες γραμμές για τους τελωνιακούς ελέγχους. όπου θα ορίσουμε κάποιες λεπτομέρειες αυτών των απαιτήσεων ασφαλείας σε στενή συνεργασία και με τις αρχές της εποπτείας αγοράς. και μετά θα ε, εκπαιδευτούν ε, οι τελωνιακοί για να εξασφαλιστεί έτσι χωρίς ε, κολλήματα συνεργασία με τις δημόσιες αρχές. Ξέρετε το θέμα αυτό της μονής θηρίδας, της μοναδικής θηρίδας, ότι πρόκειται να υπάρξει μία μοναδική θηρίδα για τους εμπόρους που να μπορούν να κάνουν ό,τι χρειάζεται για τα τελωνία, η οργία, εποπτεία και φυτογενομική εποπτεία και ούτω καθεξής. Ε, κάνουμε λοιπόν πρόεδρο στο τομέα αυτό και αυτό οδηγεί και σε πιο στενή συνεργασία μεταξύ των αρχών εποπτείας αγοράς. Χρηματοδότηση τώρα. Δύσκολο το θέμα. Και έχετε δίκιο ότι σε ορισμενα καράτη κράτη-μέλη οι πόροι έχουν περικοπεί. Στη συναντήση μου με τους υπουργούς προσπαθώ να επιμείνω ότι με το να περικόπτουν τα κονδύλια για τα τολωνία είναι σαν αυτοπυροποβολούντο, γιατί τα τολωνία προσφέρουν και έσοδα σε ένα κράτος. Και είναι πάρα πολύ σημαντικό στο επόμενο πολυεθνές ε, οικονομικό πλαίσιο να έχουμε υπόψη μας αυτά τα προβλήματα και υπάρχει η βούληση από διάφορα κράτη-μέλη να χρησιμοποιήσουν την ε, αρχή της οικονομίας κλίμακας αναπτύσσοντας τα συστήματα ε, πληροφορικής. Γιατί αν δεν γίνει αυτό θα έχουμε 27 προγράμματα ανά την Ευρωπαϊκή Ένωση. Και εμείς θέλουμε να αναπτύξουμε κάτι σε ευρωπαϊκό επίπεδο με συνεργασία μεταξύ των κρατών μελών και να διανύμουμε μετά αυτά τα σύστηματα σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση. Αυτό θα ε, πετύχει επίσης καλύτερη αρμόνιση και ευθυγράμμιση των Ταλληνίων σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση. Και έτσι και τα κράτη-μέλη θα μπορέσουν να συμβάλλουν στα διάφορα αυτά σχέδια. Και αυτό θα μας βοηθήσει να κάνουμε τις σημαντικές οικονομίες. Ευχαριστώ, Ρε Πρόεδρος. Αυτό το θέμα των προτεραιοτήτων και της είναι κάτι που παρακολουθούμε εμείς πάρα πολύ στενά. Και θα βοηθούσε βέβαια να γνώριζε καλύτερα το κοινό το ρόλο που παίζουν τα τελωνία στην ασφάλεια της εσωτερικής αγοράς. Ο κ. Σταγιάννη, ο συνάδελφός σας, μας έχει καλέσει να πάμε μαζί του σε μια επιτόπου επίσκεψη στην Αμβέρσα. Α, όχι, στο Ρότερνταμ. Ε, σχεδόν το πέτυχα. Ε, λίγο δίπλα, τέλος πάντων. <laughs> ναι, στο Ρότερνταμ θα πάμε. Αλλά καλά θα να ρωτήσετε κι εσείς ίσως. Έχω πάει, λέει ο κύριος. Αλλά θα υπάρχει και ο τύπος σίγουρα, οι δημοσιογράφοι. Ε, θα ήταν καλό να κάνετε μια παρουσία. Τώρα ήταν η πρώτη επίσκεψη που έκανα όταν έλαβα επίτροπος για την Τελωνία. Πολλά μπορούμε να μάθουμε νομίζω. Από τον τρόπο που εφαρμόζονται και τα διάφορα μέτρα. Ο κ. Κρότσμαν έχει μια ερώτηση. Και αν η κυρία Ράπτη ή η κυρία θέλουν μια ψηρωματική ερώτηση να κάνουν, θα έχουν χρόνο. Ε, κοιτάξτε, αυτό θα να σας ρωτήσω κι εγώ. Ε, δεν μπορούμε να κάνουμε μια επιτήρηση της αγοράς, αλλά σε αυτά τα πλαίσια είναι πάρα πολύ σημαντικό το τελωνίο. Εάν δεν γίνεται κάτι τέτοιο, τι αξίζει να υιοθετούμε εμείς κάποιες ε, οδηγίες κλπ θα εισάγεται άρδιν ε, ό,τι θέλει ο καθένας εδώ στην αγορά. Υπάρχουν βέβαια ορισμένα λιμάνια, τα μείνουμε στο παράδειγμα του Ρότερδα, που ε, παραλαμβάνουν πολλά, ε, πολλές εισαγωγές προς την Ευρώπη και από εκεί διανύμεται. Και πρέπει να ελέγξουμε λοιπόν τα εξωτερικά σύνορα. Είναι κάτι παρόμοιο με τους πρόσφυγες. Λέμε θα πρέπει να βοηθήσουμε εκείνες τις χώρες Πού φτάνουν οι πολλοί ε, πρόσφυγες. Σκοπεύουμε να κάνουμε κάτι παρόμοιο και όσον αφορά τα τελωνία και την επιτήρηση αγοράς. Το Αμβούργο, το Ρότερνταμ. Σας είπα, υποδέχονται εκατομμύρια αγαθών. Και όταν μπουν τα αγαθά αυτά στην Ευρώπη, διανύμονται. Και είναι πολύ σπάλιο από εκεί και πέρα τα κράτη-μέλη και μάλιστα τα ομοσπονδιακά κρατήδια στη Γερμανία που είναι υπεύθυνα για αυτά, με την επιτήρηση τη αγορά, με την αποπτήρηση τη αγορά, κάτι βρούνε. Πού κλείεται. Θα ήταν καλό λοιπόν εκείνε οι, οι χώρε, εκείνε οι πόλει που έχουν ε, τα μεγάλα λιμάνια να μην υποχρεωθούν μόνο τους να αναλάβουν όλο το βάρος πρόσληψης ε, προσωπικού σε τεράστιο αριθμό. Υπάρχει κάτι, προβλέπετε κάτι κατανομή του βάρους στα άλλα κρατημέλη ή με τον προπολογισμό της Ένωσης. Γιατί πρέπει να μην ξεχνάμε ότι και η καλύτερη τεχνολογία δεν βοηθά σε τίποτα αν δεν υπάρχουν και τα άτομα που την καλύπτουν και τη χειρίζονται. Well, of course, uh, Φυσικά δεν θέλω σήμερα να προδικάσω συζητήσεις για το επόμενο πολιετές ε, ε, οικονομικό πλαίσιο. Το Κολέγιο των Επιτρόπων εργάζεται αόκνος για το θέμα αυτό, αλλά δεν είναι ακόμα ώρα. Όταν συζητούμε για τα μελλοντικά τελωνία, και βλέποντας την γεωγραφική κατάσταση και κατανομή είναι γεγονός και είναι σαφές ότι λόγω της γεωγραφικής τους θέσης κάποιες χώρες οπωσδήποτε έχουν πολύ βαρύτερο άκθος από ό,τι άλλες όσον αφορά την προστασία των τελωνίων της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Με συμπάθεια βλέπω λοιπόν αυτήν την προσέγγιση όσον αφορά το πρόγραμμα των μελλοντικών τελωνίων. Και βεβαίως θα πρέπει να συζητηθεί το θέμα αυτό με τα συμβαλόμενα μέρη, με τους ενδιαφερόμενους, ε, με τα κράτη, με το κοινοβούλιο. Είναι γεγονός πάντως ότι υπάρχουν λιμένες που ε, έχουν μεγάλο βάρος. Έχουμε επίσης ανατολικά σύνορα τα οποία μπορεί να έχουν πάρα πολύ μεγάλο βάρος και πάρα πολύ μεγάλη πίεση γιατί είναι τα εξωτερικά σύνορα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Φυσικά θα δουλέψουμε ε, όσον αφορά την προστασία των ανατολικών συνόρων από προγράμμα, μέσα από προγράμματα για την καταπολέμηση ε, του λαθρεμπορίου κτλ. Ε, καταλαβαίνω ότι λέτε και συμφωνώ ότι η γεωγραφική θέση μπορεί να σημαίνει μεγαλύτερο βάρος τελική ερώτηση ε, από την ε, Αντιπρόεδρό μας. Κύριε Επίτροπε, θα ήθελα να σας ευχηθώ καλό κουράγιο σε σχέση με όλα αυτά που μας είπατε, γιατί σας, σας περιμένουν πολύ ζωηρές συζητήσεις με τα κράτη-μέλη. Ελπίζω ότι σε αυτό το, στον τομέα η ελληνική θα δουλέψει καλύτερα από ό,τι έχει δουλέψει σε κάποιους άλλους τομείς. Ε, εν πάση περιπτώσει, εγώ θα ήθελα να θέσω ένα ερώτημα όσον αφορά το πρώτο σημείο του νομοθετικού σας προγράμματος, κυρίως δε την κατα πολέμηση της παραχάραξης, απομίμησης κυρίως γαλλινικών ε, ε, φαρμάκων και ψεύτικων φαρμάκων. Και θα ήθελα να μου πείτε πώς μπορείτε να δουλέψετε, να συνεργαστείτε με άλλους επιτρόπους, κυρίως για να καταπολεμήσετε αυτήν την πλημμυρίδα, αυτή τη μεγάλη πληγή των παραχαραγμένων φαρμάκων στο ίντερνετ. Ε, γιατί πραγματικά δεν είναι μόνο σε εμά και σε άλλες υπήρους βλέπουμε ότι υπάρχει μεγάλη πληγή λόγω αυτών των παραποιημένων φαρμάκων. Απάντηση. Ένα σημαντικό τμήμα της ε, πρότασης για την προστασία των τελωνίων σχετίζεται με το θέμα αυτό. Και όταν μιλάμε για πωλήσει στο διαδίκτυο, ξέρουμε ότι ένα μεγάλο μέρος αφορά στα φάρμακα, αλλά βεβαίως και άλλα προϊόντα. Ξέρουμε ότι υπάρχει διακίνηση και τέτοιων προϊόντων και από αεροδρόμια και κλπ. Πάντως, θέλουμε να λύσουμε το πρόβλημα αυτό μέσα από πιο απλουστευμένες διαδικασίες για την, ε, μέσα από την καταστροφή ε, των κατασχεμένων ποσοτήτων και προτείνουμε ας πούμε να κατάσχονται όλες, όλα τα ύποπτα εμπορεύματα, είτε είναι, είτε είναι ε, ε, φάρμακα, είτε είναι άλλα είδη, και αμέσως να ξεκινάει η διαδικασία ε, αυτού που προσπάθησε, κατά αυτού που προσπάθησε να εισάγει αυτά τα αγαθά και αμέσως να καταστρέφονται ε, αυτά τα κατασχεμένα προϊόντα. Δηλαδή απλουστευμένες γρήγορες διαδικασίες έτσι ώστε τα τελωνία άμεσα να αντιμετωπίζουν τέτοιες καταστάσεις. Και βεβαίω πρέπει να σας πω ότι εμείς έχουμε πολύ μιλήσει και εξακολουθούμε να συζητούμε με τους ε, ενδιαφερόμενους... και ε, συζητούμε πάντα για τέτοιου είδους καταστάσεις, ε, για παραποιημένα προϊόντα, παραχαραγμένα φάρμακα ε, που ξέρουμε ότι πλημμυρίζουν τις αγορές μας, την αγορά της Ευρωπαϊκής Ένωσης. We uh, intend to address this subject. Ταχύτητα λοιπόν και απλούστευτη έτσι ώστε να αντιμετωπίσουμε το πρόβλημα αυτό. Θέλει κάποιος καμία τελευταία ερώτηση? Όχι. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ κύριε Επίτροπε που ήρθατε. Νομίζω ότι ήταν ε, πραγματικά έγκαιρη και πολύτιμη η ανταλλαγή απόψεων που είχαμε μαζί σας. Ε, κατανοούμε βεβαίως και την μεγάλη ε, σχέση που έχει η δουλειά σας με την εννέα αγορά. Γιατί όπως είπε και η κυρία Φανιμία προηγουμένως, ε, η, αυτού του είδους η προώθηση παραποιημένων προϊόντων, φαρμάκων κλπ. κλπ πραγματικά είναι μεγάλη απειλή για την εννέα αγορά. Ο κύριος Κρότσμαν πολύ σωστά έκανε το σχόλιο του. Δηλαδή το θέμα είναι και πώς θα χρησιμοποιήσουμε τη, τα περιφερειακά ταμεία έτσι ώστε να έχουμε μια πραγματική και ε, έγκαιρη ανάπτυξη. Ε, να ενθαρρύνουμε τις, ε, τους εμπλεκόμενους φορείς, τις επιχειρήσεις, τις εταιρείες να συμμετάσχουν στις νέες διαδικασίες να ευαισθητοποιήσουμε τον κόσμο. Και βεβαίως πολλή, πολλή δουλειά μας περιμένει ε, όσον αφορά την ε, στρατηγική ε, και χαίρομαι που πολύ συχνά έχουμε μέλη του γραφείου σας εδώ έτσι ώστε να έχουμε και ανταλλαγή απόψεων και να υπάρχει έτσι μια διαλειτουργικότητα μεταξύ μας. Οπωσδήποτε, οπωσδήποτε και εμείς από τη δικιά μας πλευρά θα κάνουμε ό,τι μπορούμε έτσι ώστε τελικά να μπορέσουμε έγκαιρα να δώσουμε την νομοθεσία που χρειάζεται. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για μια ακόμα φορά που είστε μαζί μας. Ο Επίτροπος Σεμέτα, ευχαριστώ πολύ για τα θέματα που θίξατε, για τις ερωτήσεις που μου υποβάλλατε. Προσβλέπω στην συνεργασία μας και χαίρομαι που λέτε κι εσείς ε, ότι, ότι ε, συζητούμε και συνεργαζόμαστε στενά όσον αφορά τα δικαιώματα για την πνευματική ιδιοκτησία. Ε, συζητούμε βεβαίως και με τον συναδελφό μου τον Επίτροπο Μπαρνιέ Στενή συνεργασία λοιπόν, στενή συνεργασία η οποία πιστεύω ότι τελικά θα αποβεί απολύτως εποφελής ε, και θα ε, παραγάγει καρπούς. Ευχαριστώ. Uh, so we'll have a until... Ε, θα σταματήσουμε μέχρι τις 4, 5 λεπτάκια και να πάρουν θέση και στο Προεδρείο όσοι θα πρέπει να διευθύνουν το σεμινάριο.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 Uh, um, και κύριοι, καλωσορίζω uh, όσους ήρθαν στην ειδική συνεδρίαση του απογεύματος uh, για την αμοιβαία αξιολόγηση και την οδηγία υπηρεσιών. Ξέρετε πολύ καλά ότι η οδηγία αυτή Ε, απασχόλησα από το 2004 μέχρι το 2009 την Επιτροπή μας. Και η διαδικασία αμοιβαία αξιολόγησης είναι κάτι το νέο, μια νέα διαδικασία σημαντική για την υλοποίηση της οδηγίας για τις υπηρεσίες και για να αντιμετωπίσει μερικά από τα εμπόδια τα διασυνοριακά. Γι' αυτό αποφασίσαμε να έχουμε μια έκθεση ε, και μια ανάλυση και χαίρομαι ε, που η ε, Μαλγκορζάτα Χάνσλικ είναι εδώ στο βήμα, είναι η συγγήτριά μας, είναι μια πολιτική πρωτοβουλία της Επιτροπής για να μπορούμε να έχουμε μια πλήρη συζήτηση σχετικά με το θέμα αυτό. Χαίρομαι που έχουμε εδώ διάφορους εμπειρογνώμονες που θα μας μιλήσουν για το θέμα και θα έλεγα ότι η κυρία Χάνσλικ επίσης ήταν από τους βασικούς πρωταγωνιστές, ούτω ώστε να περάσει η οδηγία για τις υπηρεσίες. Ήταν πολύ δραστήριο μέλος της Επιτροπής και ασχολήθηκε με όλη την διαδικασία υιοθέτηση της οδηγίας για τις υπηρεσίες. Ήταν μια μεγάλη εμπειρία άνευ προηγουμένου. Και ξέρω ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ε, αποδίδει ιδιαίτερη σημασία και ο κύριος Μπαρνιέ ε, έκανε πάρα πολλές επισκέψεις ε, που αποδεικνύουν το ενδιαφέρον του. Και θα επισκεφθεί σε όλα τα 27 κράτη-μέλη τις ομάδες που ασχολούνται με την υλοποίηση της οδηγίας. Ε, και ξέρω ότι αυτό ενδιαφέρει πάρα πολλούς εμπλεκόμενους, είναι πάρα πολύ λοιπόν ενθαρρυντικό το ότι μπορούμε να εξετάσουμε το θέμα αυτό λεπτομέρως. Θα ήθελα να σας παρουσιάσω, ε, πρώτα απ' όλα να παρουσιάσουμε ε, μια, ένα, έγγραφο για την αξιολόγηση που παραγγείλαμε, που ζητήσαμε. Έχουμε τον κύριο Ζωφραζέ και ο κύριο, και ο κύριος Μισάρ που θα μας παρουσιάσουν ε, το κείμενο αυτό και μετά θα τεθούν ορισμένες ερωτήσεις και μετά θα έχουμε μια ακρόαση, αλλά διάφοροι τους οποίους προσκαλέσαμε είναι από την Ανατολική και Βόρεια Ευρώπη και δεν μπόρεσαν να έρθουν λόγω της διακοπής των ε, πτήσεων ε, σήμερα Πάντως ε, θα έχουμε νομίζω μια πολύ χρήσιμη ημέρα ε, και θα μας στείλουν ε, τις παρουσιάσεις τους αργότερα. Θα, θέλαμε, θα αρχίσουμε με μια παρουσίαση της μελέτης. Ο, ο καθηγητής Βάζε θα μιλήσει πρώτος. Ε, βεβαίως θα μεταδοθεί για του διαδικτύου αυτή ε, η παρουσίαση και επίσης θα εμφανιστούν και οι διαφάνειές σας στο διαδίκτυο. Θα μπορέσουν όλοι να σας δουν, να δουν τις διαφάνειές σας. Ελπίζω ότι θα μπορέσουν επίσης ε, ε, δια, ηλεκτρονικά να έρθουν σε επαφή μαζί μας. Ο καθηγητής κ. Μπερζέ έχει τον λόγο. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι μέλη του Κοινοβουλίου εξ ονόματος των εθνικών ευρωπαϊκών οργάνων έχω την χαρά να παρουσιάσω μία εργασία για ένα θέμα που γνωρίζετε καλά, την Οδηγία 126. Το κείμενο παρουσιάζεται ως ένα κείμενο πλαίσιο, το οποίο έχει με κάποια αμφισημία, διότι προσπαθεί να κάνει μια παιδαγωγική εργασία για την νομολογία του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου για την ελευθερία εγκατάστασης και την ελεύθερη παροχή υπηρεσιών από τη δημιουργία των διαφόρων ευρωπαϊκών κοινοτήτων και ταυτόχρονα το κείμενο αυτό προσπαθεί να καινοτομήσει, να βελτιώσει τις δυνατότητες της εσωτερικής αγοράς. Στο πλαίσιο αυτών των βελτιώσεων έγινε μια πρόταση ε, και περιελήφθηκε στην οδηγία να υπάρξει ένα πλαίσιο αμοιβαία αξιολόγησης που ρυθμίζεται από ένα άρθρο, το άρθρο 39 της οδηγίας. Αυτή η διαδικασία αμοιβαία ε, αξιολόγησης έχει ως πλαίσιο ε, την οδηγία, την πρώτη εμπειρία στην Ευρωπαϊκή Ένωση και υπάρχουν και άλλες εμπειρίες στο Συμβούλιο της Ευρώπης και σε αυτήν την διάταξη του άρθρου 39 έχουμε την διαδικασία αμοιβαία αξιολόγησης για τρεις βασικές ερωτήσεις της οδηγίας, το θέμα των, της προηγούμενης αδειοδότησης, τις απαιτήσει ε, γενικού ε, συμφέροντος ε, που πρέπει να αξιολογηθούν στα κράτη-μέλη στα πλαίσια της ελευθερίας εγκατάστασης, ελεύθερης παροχής υπηρεσιών και το θέμα των πολυκλαδικών δραστηριοτήτων. Αυτά τα τρία βασικά θέματα έχουν κάτι κοινό, χαρακτηρίζουν τομείς όπου τα κράτη-μέλη συμμετέχουν με τα θεσμικά όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης στην υλοποίηση της εσωτερικής αγοράς. Γιατί? Διότι τα κράτη διατηρούν ένα περιθώριο εκτίμησης, ακόμη και αν αυτό το περιθώριο ασκείται κάτω από τον έλεγχο των, βάσει των διατάξεων της συνθήκης. Η διαδικασία αμοιβαία αξιολόγηση αυτή καθεαυτή προσδιορίζεται σε μια από τις αιτιολογικές σκέψεις της οδηγίας την 74 που περιγράφει τρία στάδια και θα δούμε ότι είναι κυρίως το δεύτερο στάδιο που μας ενδιαφέρει εδώ. Στο πρώτο στάδιο ζητείται από τα κράτη να κάνουν μια εργασία αυτοαξιολόγησης. Δεν βρισκόμαστε ακόμα στο στάδιο αμοιβαία αξιολόγησης. Κάθε ε, κράτος έχει την οδηγία και πρέπει να την ε, μεταφέρει στο εθνικό δίκαιο και κάνει μια ενδοσκόπηση κατά κάποιο τρόπο ε, για να δει με στον, στις ρυθμίσεις τις εθνικές τι τροποποιήσεις πρέπει να κάνει για να μεταφερθεί καλά η οδηγία. Έχουμε λοιπόν τα τρία αυτά θέματα ε, το θέμα της, ε, των αδειών, των προγενεστέρων, ε, της της απαιτήσει για αξιολόγηση και τις πολυκλαδικές δραστηριότητες, πρέπει κανείς να δει τις ρυθμίσεις, τους κανονισμούς, τους εθνικούς που ενδεχομένως θα μπορούν να έρθουν σε σύγκρουση με την οδηγία η οποία περιλαμβάνει τις αρχές της συνθήκης, συνθήκης ως προς την εσωτερική αγορά. Μετά από αυτή την πρώτη φάση αυτοαξιολόγησης, τα κράτη πρέπει να κοινοποιήσουν στα άλλα κράτη-μέλη την εργασία που έχουν κάνει, ούτω ώστε τα άλλα κράτη-μέλη να αντιδράσουν με τη σειρά τους σε αυτήν την εργασία αυτοαξιολόγησης κάθε κράτους μέλους. Και εδώ παρεμβαίνει με τρόπο αυστηρό η αμοιβαία αξιολόγηση. Κάθε κράτος καλείται να ακούσει και να δώσει ενδεχομένως τις εντυπώσεις του σε σχέση με την εργασία απογραφής που έκαναν τα άλλα κράτη-μέλη για να δουν αν υπάρχουν δυσκολίες. Και το τρίτο στάδιο περιγράφει πάντοτε ε, στο 74 της ε, οδηγίας είναι μια ε, συνθετική εργασία της Επιτροπής που αποτέλεσε αντικείμενο μιας μεταγενέστερης ανακοίνωσης. Έχουμε λοιπόν την φάση αυτοαξιολόγησης που είναι μια φάση που προηγήθηκε της προθεσμίας μεταφοράς της οδηγίας που ήταν 28 Δεκεμβρίου 2009, την φάση αμοιβαία αξιολόγησης που ήταν χοντρικά το έτος 2010 και είχαμε, έχουμε την ε, την ε, εργασία, την συγκεφαλαιοτική της Επιτροπής. Η αμοιβαία αξιολόγηση είναι συνεπώς μια πρωτότυπη ε, διαδικασία που δεν έχει προηγούμενο και το ε, θέμα που μας απασχολεί σήμερα είναι ποιες είναι οι μέθοδοι που ακολουθήθηκαν και ποιες είναι τα διδάγματα που μπορούμε να αντλήσουμε από αυτή την πρώτη εμπειρία. Ως προς τη μέθοδο δίνω τον λόγο στον συναδελφό μου, τον καθηγητή Φρεντερίκ Λεπλά. Σχετικά με τη μεθοδολογία που χρησιμοποιήθηκε από την Επιτροπή, το μόνο κείμενο το κείμενο της οδηγίας αποτέλεσε αντικείμενο ερμηνείας για να θεσπιστεί αυτή η διαδικασία αμοιβαία αξιολόγησης. Γίνεται σε τρία στάδια, όπως είπαμε, αυτοαξιολόγηση από τα κράτη-μέλη. Αυτό που είναι σημαντικό είναι ότι πέραν από την ανακοίνωση των εθνικών μέτρων μεταφοράς της οδηγίας κάθε κράτος μέλος έκανε μια συγκεφαλαιωτική έκθεση που εξηγεί στα άλλα κράτη-μέλη την εργασία που είχε γίνει για την ε, μεταφορά στο εθνικό δίκαιο της οδηγίας. Το δεύτερο στάδιο είναι ίσως ε, το πιο σημαντικό είναι μια εργασία που έγινε υπό clusters, δηλαδή συστάδων. Ε, δηλαδή τα κράτη-μέλη συνεδρίασαν σε περιορισμένες ομάδες για να συζητήσουν για τον τρόπο που είχαν μεταφέρει την οδηγία. Σε μια τρίτο στάδιο, με μια βαρύτερη διαδικασία, ήταν η συγκέντρωση σε ολομέλεια με το σύνολο των 27 κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ποιος ανέλαβε τη διαδικασία. Η διαδικασία αμοιβαία αξιολόγησης είναι κάτι το πρωτότυπο διότι αντιστράφηκαν οι ρόλοι. Είναι βασικά τα κράτη-μέλη τα οποία πήραν, έλαβαν το λόγο, που πήραν την πρωτοβουλία των συζητήσεων. Δεν είναι η Επιτροπή που επέλεξε και προσανατόλισε την συζήτηση μεταξύ των κρατών μελών. Είναι λοιπόν μια διαδικασία που ξεκινάει από τα κράτη-μέλη και καταλήγει στην Κομισιόν και όχι το αντίστροφο. Πρέπει να παρατηρήσουμε ότι οι σημαντικοί πόροι χρησιμοποιήθηκαν από τα κράτη-μέλη ε, για, για όλες αυτές τις συναντήσεις. Ως προς αυτό είναι σημαντικό, όπως αναφέρθηκε πριν από λίγο, ότι υπήρξαν πολλά στάδια η μεταφορά της οδηγίας και μετά η διαδικασία αμοιβαία αξιολόγησης και μόνο ε, με βάση της εργασίας αυτής σε κλάστερ, σε συστάδες, μπορούμε να μιλήσουμε ε, για μια πρωτότυπη διαδικασία. Δηλαδή, ε, τον ε, περιορισμό της ομάδος ε, για να προσδιοριστεί καλύτερα και λεπτομερέστερα αυτή η εργασία που ανέλαβαν τα κράτη-μέλη. Βεβαίω, ποια κράτη ήταν, πρόκειται για την δομή του κράτους που έχει σημασία, αν είναι συγκεντρωτικό κράτος ή αποκεντρωμένο. Τώρα θα πρέπει να δούμε εάν η διαδικασία αυτή είναι νέα, εάν είναι πρωτότυπη, μήπως υπάρχουν άλλα παραδείγματα σε άλλες οδηγίες. Αναμφισβήτητα, η αμοιβαία αξιολόγηση είναι μια πρωτότυπη διαδικασία που έχει ειδικά σχεδιαστεί και θεσπιστεί για την οδηγία για τις υπηρεσίες και στους τομείς όπου τα κράτη-μέλη είχαν ε, ένα μεγάλο περιθώριο εκτίμησης. Βεβαίως υπάρχουν μερικά παραδείγματα, κυρίως στο Συμβούλιο της Ευρώπης, αλλά πρέπει να συγκρίνουμε με τις άλλες διαδικασίες βάση του ευρωπαϊκού δικαίου. Είναι σύνηθες σε σχέση με άλλες κοινοποιήσεις που υπάρχουν, ε, είναι, πρέπει να, τα κράτη-μέλη να ανακοινώνουν στην Κομισιόν τα μέτρα μεταφοράς της οδηγίας που ε, σκέπτονται και που θα χρησιμοποιήσουν σε τομείς που καλύπτονται από μια οδηγία. Έχουμε παραδείγματα ε, κοινοποίησης, αλλά εδώ η διαδικασία αμοιβαίας αξιολόγησης είναι διαφορετική, διότι αρχίζει αφού τα ε, μέτρα ε, κοινοποίησης, έχουν, ε, τα μέσα κοινοποίησης έχουν ανακοινωθεί στην Κομισιόν. Προς την ίδια τη διαδικασία θα πρέπει να δούμε τα βασικά διδάγματα που μπορούμε να αντλήσουμε βάσει της μελέτης. Ποια είναι τα βασικά διδάγματα και συμπεράσματα. Η μελέτη ε, μας, οδήγησε να ρωτήσουμε τους εκπροσώπους των κρατών μελών ε, που συμμετείχαν στην ε, διαδικασία, όπως και την Κομισιόν, για να προσπαθήσουμε να εξαγάγουμε τα διάφορα στοιχεία και συμπεράσματα από αυτές τις εμπειρίες. Πρώτα απ' όλα, η θεώρηση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής εκφράστηκε σε μια ανακοίνωση, όπως το είπαμε. Δεν θέλω. πήραμε σε διάφορες συνεντεύξεις με την Κομισιό προκύπτει ότι πρόκειται για ένα μέσο χρήσιμο, Ερμηνεύοντας τις ανταλλαγές που είχαμε με την Κομισιό, μας, φαίνεται ότι χωρίς αυτή τη διαδικασία αμοιβαίας αξιολόγησης θα ήταν πολύ πιο δύσκολο στην Κομισιό να κατανοήσει την εμβέλεια της εργασίας που είχαν κάνει τα κράτη-μέλη. Δεκάδε χιλιάδε μέτρα μεταφορά κοινοποιήθηκαν στην Κομισιό και οι εκθέσεις που έγιναν από τα κράτη-μέλη επέτρεψαν ε, ανταλλαγές μεταξύ τους, αμοιβαία κατανόηση σχετικά με την ε, μεταφορά στο εθνικό δίκαιο, αλλά όταν η Κομισιό παρακολουθούσε αυτές τις ε, συγκεντρώσεις μπορούσε να καταλάβει ένα σημαντικό αριθμό μέτρων που χρησιμοποιήθηκαν. Αυτό που είναι ουσιώδες κατά τη γνώμη μας είναι ότι αυτή η διαδικασία αμοιβαία αξιολόγησης δεν στρέφεται μόνο προς το παρελθόν. Η Κομισιόν ήδη ανέφερε ότι αυτή η διαδικασία όπου είχε ακούσει τα κράτη-μέλη, σκεφτόταν να χρησιμοποιήσει την εργασία που έγινε για να εμβαθύνει Ε, στο θέμα της άρσης των εμποδίων στην εσωτερική αγορά. Τώρα, όσον αφορά ε, στην εμπειρία των κρατών μελών. Πραγματοποίησαμε μια μελέτη, μια έρευνα με γενικό τρόπο τα κράτη-μέλη γενικά είναι πολύ ικανοποιημένα από αυτή τη διαδικασία αμοιβαίας αξιολόγησης. Υπάρχουν βεβαίως και κριτικές, αλλά γενικά τα κράτη-μέλη όλα θεώρησαν ότι αυτή η διαδικασία αμοιβαία αξιολόγηση ήταν ιδιαίτερα ενδιαφέρουσα και τους επέτρεψε να κατανοήσουν καλύτερα και να ανταλλάξουν μεταξύ τους ιδέες και να έχουν μια καλύτερη εικόνα της εσωτερικής αγοράς ε, ερχόμενοι αντιμέτωποι με την εμπειρία των άλλων κρατών μελών. Υπήρξαν βεβαίως κριτικές η Αυστρία ε, εξέφρασε επιφυλάξεις, αλλά πρέπει να παρατηρήσουμε ότι ακόμα και οι χώρες που εξέφρασαν τις περισσότερες κριτικές δεν ήταν αρνητικές, ε, δεν ε, εγκατέλειψαν το παιχνίδι αυτό. Απλώς σκέφτηκαν ότι ήταν καλύτερα να συναντήσουν χώρες που βρίσκονται πιο κοντά, η Αυστρία με τη Γερμανία το χάρη, για να δουν μαζί τις δυσκολίες. Δεν ήταν μια άρνηση μιας κοινή ανταλλαγής, αλλά παραδείγματος χάρη η χώρα αυτή θεώρησε ότι θα ήταν πιο αποτελεσματικό να ακολουθήσει μια άλλη μέθοδο και να μην συμμετέχει στις ολομέλειες που είχαν πιο περιορισμένα αποτελέσματα από την, τις περιορισμένες ομάδες. Έχουμε λοιπόν ένα feedback αρκετά θετικό από τα κράτη-μέλη για αυτή τη διαδικασία. Όπως επισημάναμε, ακόμα και οι χώρες που εξέφρασαν κριτικές ε, συναντήθηκαν ξεχωριστά για να προσπαθήσουν να εμβαθύνουν σε αυτή την εργασία μεταφοράς στο εθνικό δίκαιο ποια είναι, ποια είναι η εικόνα των κρατών μελών, η θεώρηση των κρατών μελών. Λοιπόν, πρέπει να δούμε τώρα τι γίνεται με τα εμπλεκόμενα μέρη, του stakeholders και τη συμβολή τους σε αυτή την εργασία αμοιβαία αξιολόγησης. Τα ενδιαφερόμενα εμπλεκόμενα άτομα δεν συνδέθηκαν άμεσα ε, με τις ε, συνεδριάσεις μεταξύ των κρατών μελών. Ε, δώσανε τη γνώμη τους ε, κυρίως για την μεταφορά της οδηγίας και κυρίως σε εθνικό επίπεδο. Μετά την εργασία αμοιβαία αξιολόγησης, η Κομισιό ε, συμβουλεύτηκε ηλεκτρονικά τα διάφορα ενδιαφερόμενα μέρη και άτομα. Στις διάφορες ε, συγκεντρώσεις συστάδες, σε κλάστερς ή σε ολομέλειες, μόνο τα κράτη-μέλη ήταν παρόντα και πάρα πολλέ λίγες πληροφορίες δόθηκαν και τα ενδιαφερόμενα άτομα δεν μπόρεσαν να παρακολουθήσουν την εργασία αμοιβαία αξιολόγηση και το αντικείμενο των ανταλλαγών. Από την άποψη αυτή αναμφισβήτητα υπήρξε πολύ λίγη διαφάνεια, πράγμα που εξηγεί τις κριτικές που διατυπώθηκαν, ένα μέρος των κριτικών. Μόνο η ανακοίνωση της Επιτροπής δίνει μια ιδέα της εργασίας που έχει γίνει. Τώρα πρέπει να δούμε τις συνέπειες αυτής της εργασίας αμοιβαίας αξιολόγησης. Για να κατανοήσουμε καλύτερα θα πρέπει να έχουμε υπόψη ότι η αμοιβαία αξιολόγηση έγινε μετά την μεταφορά της οδηγίας. Μετά, ε, αφού εξέπνευσε η προθεσμία, τα κράτη-μέλη συναντήθηκαν μεταξύ τους για να εξετάσουν, να κατανοήσουν τι είχαν κάνει τα άλλα κράτη-μέλη. Το... Τέθηκε το ερώτημα στα κράτη-μέλη του εάν η αμοιβαία αξιολόγηση είχε επηρεάσει την επιλογή τους ως προς την οδηγία για τις υπηρεσίες. Στην πλειονότητά τους τα κράτη-μέλη θεώρησαν ότι αυτή ήταν η περίπτωση, ότι έτσι είχε γίνει. Πέραν από αυτό το ερωτηματολόγιο πρέπει να καταλάβουμε ότι κανένα συγκεκριμένο παράδειγμα δεν μας δόθηκε για άμεση επίδραση της διαδικασίας αμοιβαίας αξιολόγησης πάνω στις επιλογές που είχαν γίνει σχετικά με αυτήν την οδηγία για τις υπηρεσίες. Άλλη μια φορά ήταν πολύ αργά για να επανέλθουμε στο θέμα της ε, μεταφοράς το, το κείμενο το εθνικό είχε υιοθετηθεί ή υιοθετεί το τότε, συνεπώς η εργασία προβληματισμού δεν μπορεί να θεωρηθεί ως μέσο διευκόλυνσης μιας καλύτερης μεταφοράς της οδηγίας. Το πραγματικό συγκεκριμένο αποτέλεσμα της διαδικασίας αμοιβαίας αξιολόγησης είναι η δυνατότητα μιας καλύτερης κατανόησης της εργασίας που έγινε σε κάθε κράτος μέλος. Η Επιτροπή το επεσήμανε στην ανακοίνωσή της, αλλά η έρευνα που έγινε το δείχνει ακόμη σαφέστερα. Αναμφισβήτητα υπήρξε μια πνοή ευρωπαϊκή στις εθνικές διοικήσεις που συμμετείχαν σε αυτή τη διαδικασία αμοιβαία αξιολόγησης. Ο καθένας μπόρεσε να εντάξει καλύτερα με συγκεκριμένο παράδειγμα την οδηγία την ευρωπαϊκή, βλέποντας τι έχουν κάνει οι άλλοι. Υπήρξε, λοιπόν, υπήρξαν λοιπόν συνέπειες αυτής της διαδικασίας αμοιβαίας αξιολόγησης με μια καλύτερη ένταξη του ευρωπαϊκού συμφέροντος στις εθνικές διοικητικές αρχές και έτσι μπορούμε να διαιρετηθούμε για την μονιμότητα των ανταλλαγών μεταξύ εθνικών ε, διοικήσεων που προκλήθηκε από αυτήν τη διαδικασία αμοιβαία αξιολόγησης. Ε, επίσης το θέμα του λόγου ανάμεσα στο κόστος και στα ωφέλη είχε σημασία. Τα περισσότερα κράτη-μέλη θεώρησαν, η πλειονότητά τους θεώρησε ότι τα ωφέλη ήταν ανώτερα από το κόστος αλλά δεν είναι βέβαιο ότι η απάντηση των εθνικών δικήσεων ήταν, ε, ήταν βάσιμη πάντοτε, διότι δεν ξέρουν πολύ καλά το κόστος και τα ωφέλη. Έχουμε πολύ λίγα συγκεκριμένα αποτελέσματα μετά τη μεταφορά. Υπάρχουν πιο άειλα αποτελέσματα, καλύτερη κατανόηση εργασίας που έγινε από άλλες εθνικές αρχές. Αυτή η αξιολόγηση είναι πρόορη. Τα πάντα θα εξαρτηθούν από το τι θα κάνει η Κομισιό από την εργασία που έγινε σε αυτήν την διαδικασία αμοιβαία αξιολόγηση. Αν με τα μελλοντικά μέτρα η Κομισιό αποδείξει ότι η διαδικασία αυτή έχει συγκεκριμένα αποτελέσματα στις προτάσεις, τότε αναμφισβήτητα η διαδικασία υπήρξε χρήσιμη ακόμη και μόνο αν έχει επιτρέψει στην Κομισιό να δει τις επιπτώσεις στην εσωτερική αγορά και να βελτιώσει την εργασία για την εξάλληψη των εμποδίων. Αν αυτή η εργασία μείνει χωρίς επιπτώσεις, αν δεν λάβει καμιά πρωτοβουλία η Κομισιόν, θα πρέπει να είμαστε πιο επιφυλεκτικοί ως προς την σύγκριση του κόστους και της ωφέλειας. Είναι πρόωρο σήμερα να μπορέσουμε να αποφανθούμε κατηγορηματικά για την σχέση μεταξύ κόστους και ωφέλους αυτής της διαδικασίας. Η μπάλα βρίσκεται στα χέρια της Κομισιό και μπορούμε να συμπεράνουμε ότι υπήρξαν δύο προσεγγίσεις της διαδικασίας αμοιβαία αξιολόγησης. Σε μια πρώτη προσέγγιση η διαδικασία είναι μια ανταλλαγή μετά τη μεταφορά της οδηγίας που έχει λίγο αντίκτυπο ε, υπήρξε καλύτερη κατανόηση, αλλά είναι δύσκολο να αιτιολογηθεί ο αντίκτυπος με το, τις δαπάνες που χρειάστηκαν και μια δεύτερη προσέγγιση της Κομισιόν και η δική μας. Η διαδικασία δεν στρέφεται προς το παρελθόν, αλλά προς ε, τα μέτρα που έχουν ήδη ληφθεί για την μεταφορά και στρέφεται προς το μέλλον της εσωτερικής αγοράς. Η διαδικασία αυτή είναι το σημείο κίνησης μιας νέας εργασίας που πρέπει να κάνει η Κομισιό, εργασία που κατέστη δυνατή από τις ανταλλαγές που έλαβαν χώρα μεταξύ των κρατών μελών. Ε, θα αφήσω τον συνάδελφο Μπερζέ να συμπεράνει για τα διδάγματα που μπορούμε να αντλήσουμε από αυτή τη διαδικασία. Όσον αφορά τα μαθήματα, ε, μπορούμε να αναφέρουμε δύο στοιχεία, τα οποία θα πρέπει να συγκρατήσουμε. Πρώτον, ότι υπήρχε μία αμφιβολία όσον αφορά την φιλοδοξία του προγράμματος αμοιβαίας αξιολόγησης. Ε, δηλαδή κατά πόσο θα έπρεπε να δούμε το παρελθόν, εάν η μεταφορά έγινε σωστά ή όχι, ή εάν θα έπρεπε να βλέπουμε, να δούμε προς το μέλλον, να έχουμε ένα εργαλείο δηλαδή ε, εγγεγραμμένο στην προοπτική του μέλλοντος. Η απάντηση σε αυτό το πρώτο ερώτημα είναι ότι ε, χωρίς να γνωρίζουμε ακόμα πλήρως ε, την εκμετάλλευση της οποίας θα τύχει η διαδικασία αμοιβαίας αξιολόγησης, διαπιστώνουμε παρόλα αυτά ότι πρόκειται για ένα εργαλείο στραμμένο προς το μέλλον. Πρόκειται για θέματα τα οποία δεν καλύπτονται πλήρως από την παρούσα οδηγία, πρόκειται για θέματα τα οποία είναι συζητημένα, αλλά και περίπλοκα και πολύπλοκα. Επ' αυτών ξέρουμε ότι η διαδικασία θα συνεχιστεί και επομένως ε, η διαδικασία αμοιβαίας αξιολόγησης ε, πρέπει να ε, μελετηθεί περαιτέρω. Δεύτερο ερώτημα, να, ξέρουμε, να μάθουμε, να δούμε εάν αυτή η διαδικασία αμοιβαίας, αξιολόγηση αξιολόγησης είναι αρκετή για τα κράτη και εάν είναι μια ενδιαφέρουσα διαδικασία για, το, για τα κράτη. Εδώ θα κάνω μια προσωπική αξιολόγηση οτιδήποτε σχετίζεται με την συνεργασία ανάμεσα στα κράτη, συνεργασία απαραίτητη για την δημιουργία ε, του, του ευρωπαϊκού οικοδομήματος. Ε, όλες αυτές ε, οι διαδικασίες αξιολόγησης είναι πάρα πολύ σημαντικές. Δηλαδή, οι διάφοροι οργανισμοί, υπηρεσίες κλπ. ανταλλάσσουν εμπειρίες, ανταλλάσσουν γνώμες έτσι ώστε να ορίσει η καθεμία μία περίμετρο δράσης. Βεβαίως αυτό μπορεί να μην είναι γενικευμένο παντού και σε όλους τους όμως είναι πάρα πολύ σημαντικό να σκεφτούμε ότι ε, μια ευρωπαϊκή δράση η οποία έχει επιβληθεί εκ των άνω ε, μπορεί να δημιουργήσει χώρους στους οποίους μπορούν να λειτουργήσουν και να συναντηθούν οι διάφορες υπηρεσίες. Κατά αυτή την έννοια πιστεύω ότι μπορούμε ε, να διατηρήσουμε και οφείλουμε να διατηρήσουμε το ενδιαφέρον αυτής της διαδικασίας. Ευχαριστώ πολύ. Σας ευχαριστούμε πολύ. Ζητώ συγγνώμη γιατί δεν έκανα μάλλον καλά τις, ε, την παρουσίαση των εμπειρογνωμόνων. Πάντως βλέπετε ότι πρόκειται περί των νομομαθών. Ο κύριος Μπερζέ, ο κύριος Λεπάρ έχουν ε, πραγματικά ε, ευρία πείρα όσον αφορά τα θέματα αυτά. Ε, και είναι πολύ σημαντικό να έχουμε την άποψή τους όσον αφορά αυτές τις νέες εξελίξεις. Ε, θα ήθελα πριν ανοίξω τη συζήτηση να καλωσορίσω ε, την, την εκπρόσωπο της European Work Council Ε, διότι μέσα από ε, ε, τέτοιες εμπειρίες μπορούμε να δούμε πώς έχουν τα πράγματα στο δημόσιο αλλά και στον ιδιωτικό τομέα. Εν πάση περιπτώσει, ξέρουμε ότι εσείς γνωρίζετε πώς γίνονται οι πολιτικές συζητήσεις και μπορείτε να πάρετε μέρος και στη δική μας συζήτηση. Επίσης, να καλωσορίσω την συνάδελφο κυρία Γκέπχαρτ, η οποία είναι και η συγγήτρια, για τα θέματα αυτά και έχει κάνει πολλές εκθέσεις για όλα αυτά τα θέματα ε, και είναι πολύτιμη η παρουσία της. Θα συνεχίσουμε, αλλά Ε, μπορούμε να έχουμε και κάποιες ανταλλαγές ε, απόψεων. Οπωσδήποτε οι συνάδελφοι ε, θα θέσουν ερωτήματα και θα κάνουν σχόλια σχετικά με όσα ακούσαμε. Αν θέλουν να θέσουν κάποια ερωτήματα άμεσα οι συνάδελφοι, μπορούμε τώρα να έχουμε μία σειρά ερωταπαντήσεων και μετά να συνεχίσουμε με το υπόλοιπο πάνελ και τις υπόλοιπες παρουσιάσεις. Ε, θα ήθελα τώρα να καλωσορίσω την κυρία Πάμελα Μπρόμτερ, η οποία ε, εκπροσωπεί την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Θα μιλήσετε από τη θέση σας ή θέλετε να έρθετε προς τα δω. Η κυρία Μπρόμτερ είναι επικεφαλής ε, της μονάδας που ήταν ε, υπεύθυνη για την ε, αμοιβαία αξιολόγηση και την εφαρμογή της. Συχνά είχαμε τακτικές επισκέψεις από μέλη της ομάδας της και χαιρόμαστε πάρα πολύ κυρία Μπρόμτερ που σας έχουμε μαζί μας. Όμως, θα ήθελα να, κάνω κάποιες, ε, να κάνουμε κάποιες πρώτες ε, παρατηρήσεις και επομένως ε, να καλέσω την εισηγήτριά μας κυρία Μαλγκορτζάτα Χάντζλικ να κάνει κάποιες πρώτες παρουσιάσεις. Ευχαριστώ πάρα πολύ κύριε Πρόεδρε. Είμαι πάρα πολύ ευτυχής που μπορούμε να συζητήσουμε σήμερα τα θέματα αυτά το θέμα της αμοιβαία αξιολόγησης που είναι ένα πάρα πολύ σημαντικό ε, ζήτημα και το οποίο για πρώτη φορά αναφέρεται στην οδηγία για τις υπηρεσίες. Ε, αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό για τα κράτη-μέλη και είμαι ιδιαίτερως ευτυχής επίσης. Ε, διότι η οδηγία για τις υπηρεσίες είναι κατά κάποιο τρόπο μωρό της Επιτροπής μας εδώ, της ε, ΙΜΚΟ και αυτό με χαροποιεί ιδιαίτερα. Συζητήσαμε πρόσφατα τα θέματα αυτά με την ευκαιρία της εκθέσεως Γκέπχαρτ για την ε, υλοποίηση και εφαρμογή της οδηγίας. Κυρίες και κύριοι, η αμοιβαία αξιολόγηση έχει εγγραφεί πλέον στην οδηγία και είναι σημαντικό να σημειώσει κανείς ε, ότι με αμοιβαία αξιολόγηση, μάλλον ε, δεν υπάρχει σε, όλες τις, ε, σε όλα τα της οδηγίας, αλλά αφορά την λειτουργία των επιχειρήσεων, κυρίως σε σχέση με το άρθρο 39 και ε, με, το, με τις πολυτομιακές δραστηριότητες του 15 ε, καθώς επίσης ε, και στην διασυνοριακή παροχή υπηρεσιών άρθρο 16 της οδηγίας. Σχετικά με την αμοιβαία αξιολόγηση δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι είναι κάτι πάρα πολύ σημαντικό και είναι κάτι που έχει, έχουμε συζητήσει εδώ και πάρα πολύ ε, καιρό. Ολόκληρο το 2010 συζητούσαμε το θέμα αυτό ε, και τον Ιανουάριο του 2010 η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δημοσίευσε μία έκθεση με συνοδευτικό, μία ανακοίνωση με συνοδευτικό έγγραφο σχετικά με τη διαδικασία αμοιβαίας αξιολόγησης ε, και περιέγραψε ε, δράσεις οι οποίες θα έπρεπε να ληφθούν στο εγγύς μέλλον. Και εύχομαι η εκπρόσωπος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής να μας δώσει και λεπτομέρειες για τα θέματα αυτά τα έγγραφα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής ε, είναι αυτά τα οποία ε, αποτέλεσαν τον μπούσουλα κατά κάποιο τρόπο για τις συζητήσεις που έλαβαν χώρα και στα κράτη-μέλη στη σημερινή ακρόαση ε, θέλουμε να δούμε λεπτομέρειες της ε, οργάνωσης της αμοιβαίας αξιολόγησης. και να ακούσουμε κάποιες σκέψεις οι οποίες ε, θα αποτελέσουν και έναυσμα και για τη δικιά μας περαιτέρω σκέψη όσον αφορά τα θέματα αυτά. Γι' αυτό λοιπόν χωρίσαμε το σεμινάριο το σημερινό, την ακρόαση τη σημερινή σε δύο ε, τμήματα. Ε, στο τμήμα που αφορά την πράξη για την ενιαία αγορά ε, αναφερόμαστε στην σημασία που έχει η αμοιβή αξιολόγηση για την εμβάθυνση της ιδείας και πώς μπορεί η αμοιβαία αξιολόγηση να βοηθήσει την λειτουργία της ενιαίας αγοράς. Θα ακούσουμε και εκπροσώπους της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, εκπροσώπους χωρών. Έχουμε, ε, ε, δυστυχώς ε, είχαμε πολύ περισσότερους εκπροσώπους των εργαζομένων, των εργοδοτών, που όμως δυστυχώς δεν μπορεί να είναι μαζί μας λόγω των προβλημάτων που ο πρόεδρος Χάρμπορ ανέφερε στην αρχή της συνεδρίασης. Πάντως μπορώ να σας πω και να σας διαβεβαιώσω ότι είναι αρκετέ οι χώρε οι οποίες δουλεύουν ομαδοποιημένα σε clusters ε, έτσι ώστε να ε, μεταφερθεί και να εφαρμοστεί όσο γίνεται καλύτερα η οδηγία. Η Γαλλία θα παρουσιάσει ε, και ένα πολύ ευρύ ε, φάσμα ε, εργασιών που έχουν κάνει όσον αφορά την ανάπτυξη της αμοιβαίας αξιολόγησης. Ακούσαμε επίσης και δύο έγκριτους Βέλγους που μας είπαν πολύ σημαντικά πράγματα σχετικά με την αμοιβαία αξιολόγηση. Είναι σημαντικό να ακούσουμε, ε, αλλά να προσέξουμε και να θέσουμε και εμείς ερωτήματα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ ε, για την παρουσία σας, για την παρακολούθηση ε, και πραγματικά ελπίζω ότι αφού θα έχουμε ακούσει όλο το πάνελ θα έχουμε εμβαθύνει τις γνώσεις μας όσον αφορά την διαδικασία αμοιβή αξιολόγηση. Ευχαριστώ. Πρόεδρος. Νομίζω ότι όλα αυτά που θα συζητήσουμε σήμερα το απόγευμα θα μας οδηγήσουν ε, σε εμβάθυνση των γνώσεών μας όσον αφορά την αμοιβαία αξιολόγηση. Λοιπόν, να σας πω. Έχουμε τώρα δύο στοιχεία, δύο κομμάτια. Για την επόμενη ώρα θα μιλήσουμε για την διαδικασία αμοιβαίας αξιολόγησης, εμπειρίες, αποτελέσματα και βήματα περαιτέρω. Ε, γιατί ένα από τα ζητήματα τα οποία κατεδείχθησαν και από τη δικιά μας έρευνα είναι πόσο αποτελεσματική ή ε, πόσο ε, σημαντική μπορεί να είναι η επίπτωση αμοιβαίας αξιολόγησης στην ενιαία αγορά. Επομένως, με ποιο τρόπο μπορούμε να ενδυναμώσουμε τη διαδικασία έτσι ώστε να έχει μια πραγματική, ένα πραγματικό αντίκτυπο στην ενιαία αγορά. Αυτά θα συζητήσουμε στο πρώτο κομμάτι. Και στην πράξη για την ενιαία, για αγορά τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή, η εμβία αξιολόγηση είναι ένα εργαλείο το οποίο όμω μπορεί να εφαρμοστεί και σε άλλα ε, κομμάτια τη ενιαίας αγορά. Και ε, το ερώτημα, ένα από τα ερωτήματα τα οποία προκύπτουν από την μελέτη είναι ε, τι μπορούμε να κάνουμε και πώς μπορούμε να προχωρήσουμε. Θεωρητικώς όλοι πρέπει να έχετε ένα αντίγραφο των του προγράμματος, καθώς επίσης και αντίγραφο της, του, των βιογραφικών σημειωμάτων των εμπειρογνωμόνων. Η μελέτη που είδατε και το λέω κυρίως για αυτούς που ε, παρακολουθούν μέσω διαδικτύου είναι διαθέσιμη και online επιγραμμικά και επομένως μπορείτε να την κατεβάσετε αν θέλετε. So uh, Uh, Θα έχουμε λοιπόν πρώτα την κυρία Πάμελα Μπρόμπτερ Κορέκτ μετά την, από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, την κυρία Ελέν Μασάρ από το Υπουργείο Οικονομίας της ε, Γαλλίας. Έχουμε την κυρία Άννα Βίλ Σεπαρκόφσκα, δεν είμαι σίγουρος ότι το προφέρω καλά, από το Υπουργείο Οικονομίας της Πολωνίας. Ε, είναι η αναπληρώτρια διευθύντρια του Τμήματος Ευρωπαϊκών Υποθέσεων. Έχουμε την κυρία Άννα Στραντμπακ η οποία ίσα ίσα ξέφυγε ε, από το, ε, ε, από τον του ηφαιστείου της Ισλανδίας για να προσγειωθεί στις Βρυξέλλες και την ευχαριστούμε γι' αυτό. Έχουμε την κυρία Ναταλή Ζουάν, η οποία είναι policy officer από την περιφέρεια των Βρυξελών, της πρωτεύουσας δυστυχώς ε, δεν είναι δυνατόν να έχουμε την εκπρόσωπο της Αυστρίας, την κυρία Σιμπίλ, τον κύριο μάλλον Λούκας Όμπερντόρφερ και θα έχουμε την κυρία Σιμπίλ uh, To uh, Ούτε την κυρία Σιμπίλ Κούζαθ, οι οποίοι θα, και οι δύο θα, θα υποβάλουν γραπτά τις ε, παρεμβάσεις τους. Λοιπόν, ε, κυρία Μπρόμτερ, παρακαλώ να ξεκινήσετε. Ευχαριστώ πολύ. Εγώ θα σας πω δύο λόγια από πλευρά της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τον τρόπο με τον οποίο ε, εμείς αντιμετωπίζουμε αυτήν την ε, νέα διαδικασία. Να σας πω δύο λόγια σχετικά με το περιβάλλον στο οποίο δουλέψαμε ε, πέρσι με τους εμπειρογνώμονές μας. Λοιπόν, ξεκινήσαμε να μελετούμε τις υποχρεώσεις της οδηγίας και μία από αυτές ήταν η αμοιβαία αξιολόγηση. Δεν καλύπτει το σύνολο της οδηγίας, αλλά καλύπτει κάποια ειδικά στοιχεία και κάποιες ειδικέ πρόνοιες της ε, οδηγίας. Όμως η οδηγία αφήνει ένα μεγάλο ε, περιθώριο διακριτικής ευχέρειας ε, για τα κράτη-μέλη έτσι ώστε να αντιμετωπίσουν ενδεχόμενα εμπόδια και να τα ξεπεράσουν. Κατά αυτή την έννοια ε, εδώ δεν μιλάμε για ε, διαδικασία ή εργασία μεταφορά στο εθνικό δίκαιο ε, και εργαστήκαμε και γι' αυτό, αλλά πριν από την... Αλλά η άσκηση αυτή για τη μεταφορά είναι μια διαφορετική άσκηση από την αμοιβαία αξιολόγηση. Αυτό που θέλουμε να αξιολογήσουμε είναι να δούμε πώς δούλεψαν τα κράτη μέσα στα πλαίσια των αποφάσεων που έπρεπε να λάβουν ε, στα πλαίσια των περιοθωρίων που είχαν βάσει τις ε, οδηγίες και πώς προχώρησαν με αυτή την αξιολόγηση. Η, αξιολόγηση, όπως ήδη, η αξιολόγηση όπως ήδη αναφέρθηκε ε, έπρεπε να απαντά σε κάποιες ειδικέ απαιτήσει των αξιολογητών ε, όσον αφορά την νομική ε, ισχύ αφενός αλλά και την διασυνοριακή παροχή υπηρεσιών κτλ. Οτιδήποτε προβλέπεται στην οδηγία για τις υπηρεσίες. Είχαμε ε, συγκεκριμένες προθεσμίες και χρονικά ε, όρια ε, και συγκεκριμένα έπρεπε να έχει ολοκληρωθεί η εργασία μέχρι το τέλος του 2010. Και για μας η μεγάλη πρόκληση ήταν να μπορέσουμε να αντιμετωπίσουμε, με αυτό το, να αντιμετωπίσουμε αυτό το πολύ φιλόδοξο πρόγραμμα και ας πούμε για να αναφέρω την τι απαιτήσει από πλευρά ε, κρατών μελών είχαμε 35.000 ε, ε, απαιτήσει, επομένως μεταξύ Ιανουαρίου και Οκτωβρίου 2010 μέσα σε 10 μήνες δηλαδή έπρεπε να ολοκληρώσουμε αυτές τις διαδικασίες και επιπλέον και για να κάνει ακόμα πιο περίπλοκη την διαδικασία έπρεπε να αναμειχθούν στη διαδικασία αυτή όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη έτσι ακριβώ όπω απαιτούσε η οδηγία. Με τον καλύτερο δυνατό τρόπο λοιπόν προσπαθήσαμε να αντιμετωπίσουμε αυτές τις ε, ε, υποχρεώσεις. Δουλέψαμε πολύ και βασιστήκαμε πολύ στα κράτη-μέλη. Δουλέψαμε, τα κράτη-μέλη δηλαδή οργανώθηκαν σε κλάστερ και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ήταν πάντα κοντά τους να τους βοηθήσει στην οργάνωση. Όμως είναι ορθό να πούμε ότι τελικά τα κράτη-μέλη διοίκησαν κατά κάποιο τρόπο, οδήγησαν ε, την διαδικασία μέσω των clusters και πρέπει να πω ότι αυτή η διαδικασία ήταν νέα, καινούρια. Δεν μπορούσε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να, ε, ε, ε, να υποχρεώσει τα κράτη-μέλη να οδηγηθούν στη διάρκεια της αξιολόγησης αυτής προς μία συγκεκριμένη κατεύθυνση. Τα ίδια τα κράτη-μέλη έπρεπε να οδηγήσουν τη διαδικασία, να συγκρίνουν τα συστήματα, ε, να αποφασίσουν γιατί κάποιες, ε, ε, κάποιοι περιορισμοί έπρεπε να παραμείνουν σε ορισμένα συγκεκριμένα ζητήματα ή εάν μπορούσαν να αρθούν οι περιορισμοί ή εάν μπορούσαν να υπάρξουν εναλλακτικά, εναλλακτικοί τρόποι. Άλλωστε μερικές χώρες μέλη βρήκαν εναλλακτικούς τρόπους. Ο εμπειρογνώμονας που ακούσαμε προηγουμένως ανέφερε ότι ε, δεν υπήρχε υποχρέωση να αλλάξουν τα νομικά συστήματα κάποιων χωρών οι οποίες δεν συμφωνούσαν. Αυτό είναι πολύ δύσκολο να το πούμε σήμερα και να το αξιολογήσουμε. Πάντως υπάρχουν κάποιες χώρες μέλη οι οποίες έχουν αλλάξει ε, άποψη ε, και βλέπουν ξανά λίγο πώς είναι το νομικό τους σύστημα. Ε, και εν πάση περιπτώσει αυτό αποτελεί ένα πιο θετικό βήμα από αυτό στο οποίο αναφέρθηκαν οι εμπειρογνώμονες που μόλις ακούσαμε. Η διαβούλευση των συμβαλωμένων ε, και ενδιαφερομένων μερών, και αυτό ήταν ένα σημαντικό θέμα στη διαδικασία μας, είναι πάρα πολύ δύσκολο για τους εμπλεκόμενους να εξετάσουν 35.000 ε, απαιτήσει. Ήταν απόλυτα αδύνατο από τη δικιά τους πλευρά και ήταν ε, πολύ δύσκολο να, να εμπλακούν στη διαδικασία συζήτησης μέσω κλάστερς. Τι κάναμε λοιπόν, κάναμε ε, ένα έγγραφο ε, για αυτούς, ένα είδος σύνθεσης, ένα είδος περίληψης του τι συζητείται στα κλάστερς και στην Ολομέλεια και αυτό ακριβώς το έγγραφο υποβάλαμε σε δημόσια διαβούλευση τον προηγούμενο Ιούνιο, Ιούνιο του 2010. Αφήσαμε αρκετό χρόνο για τη διαβούλευση με τα, τους εμπλεκόμενους φορείς και αυτός κατά την άποψή μας ήταν ένας τρόπος διαβούλευσης που ε, τους έδινε την δυνατότητα να εμπλακούν και να απαντήσουν χωρίς να ε, ακολουθήσουν όλα τα στάδια της διαδικασίας που θα ήταν δύσκολο και για μας και για αυτούς. Το χρονοδιάγραμμα ήταν πάρα πολύ σφιχτό βεβαίως Ακόμα και αν θέλαμε να έχουμε μεγαλύτερη εμπλοκή των διαφόρων φορέων, ο χρόνος δεν μας το επέτρεπε, ήταν πάρα πολύ δύσκολο να το κάνουμε και επομένως ακριβώς επιλέξαμε αυτήν την ε, διαδικασία διαβούλευσης. Ε, όσον αφορά τώρα ε, τα αποτελέσματα της αμοιβαίας αξιολόγησης, οι εμπειρογνώμονες είπαν ότι κοιτούμε προς το μέλλον, είναι μια προοπτική και αυτό κατά την άποψή μου είναι απολύτως ορθό. Αυτός άλλωστε ήταν και ο στόχος όλης της άσκησης και της προσπάθειας. Και στην ανακοίνωσή μας το συμπέρασμα το οποίο απορρέει κατά την άποψή μας από αυτή την άσκηση είναι ότι ε, είδαμε σε διάφορους τομείς ε, τι πρέπει να γίνει, ποιοι είναι οι περιορισμοί οι οποίοι είτε πρέπει να συνεχίσουν είτε πρέπει να αρθούν. Είναι γεγονός ότι ε, κάποιες χώρες δεν έχουν άρει ορισμένους περιορισμούς και επομένως πρέπει να συνεχίσουμε την προσπάθεια. Πρέπει να επικεντρώσουμε τώρα την δράση μας σε αυτά τα ειδικά ζητήματα τα οποία ε, αναφέραμε, ας πούμε τις ε, legal forms, ε, επίσης την συγκεκριμένες δραστηριότητες οι οποίες μπορεί να διαφέρουν από χώρα σε χώρα για τις οποίες εξακολουθούν να υπάρχουν κάποιες επιφυλάξεις. Τώρα η δουλειά μας θα πρέπει να γίνει περισσότερο σε βάθος έτσι ώστε να καταλήξουμε σε συγκεκριμένες προτάσεις. Αφού λοιπόν θα έχουμε ενδελεχέστερα και πιο εμπεριστατωμένα μελετήσει κάποιους τομείς τότε θα κάνουμε και τους ε, δεύτερους ελέγχους, ε, θα κάνουμε τους ελέγχους επιτόπου, θα έχουμε τη δυνατότητα να συνδυάσουμε εφαρμογή διαφόρων νομοθεσιών και με πολύ συγκεκριμένο τρόπο να προχωρήσουμε. Κατά αυτή την έννοια ευελπιστούμε ότι θα έχουμε συγκεκριμένα αποτελέσματα σε συνεργασία με τα κράτη-μέλη Συνεχίζουμε βεβαίως την καλή σχέση που έχουμε δημιουργήσει. Θα την συνεχίσουμε αυτήν την καλή σχέση και θα συνεχίσουμε με τους ελέγχους αποδοτικότητας και στο μέλλον. Και αυτά θέλω να πω. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Και εγώ σας ευχαριστώ. Θα έχετε την ευκαιρία να ξανεβανέσετε βέβαια όλοι αλλά είναι πάρα πολύ σημαντικό να σε ακούσουμε τώρα για να ακούσουμε εκείνους που άμεσα ασχολήθηκαν με το θέμα αυτό. Θα δώσω καταρχήν το λόγο στην κυρία Έλεν Μασάχα, που είναι, εργάζεται στο Γαλλικό Υπουργείο Οικονομικών. Παρακαλώ κυρία Μασάχα, έχετε το λόγο. Ε, καλημέρα σας και σας ευχαριστώ Πρόεδρε. Θα την ευχαριστήσω το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και την, Κομισιόν, την Επιτροπή ΕΜΚΟ για την πρόσκληση αυτή. Είναι πάρα πολύ σημαντικό να έρχεται ένα να ε, παρουσιάσει τα αποτελέσματα της διαδικασίας αμοιβαίας ε, αξιολόγησης που κοινοτοποίησε τα κράτη-μέλη επί 10 μήνες. Πάρα πολύ σημαντικό αυτό για την ε, οδηγία για τις υπηρεσίες. Η θέση της Γαλλίας είναι γενικά θετική για τη διαδικασία αυτή και η, μελέτη των κυρίων Μπεζό και Λεπλά ανεκατοπρίζει απόλυτα αυτή την άποψή μας. Είναι ένα καινοτομικό μέσο γιατί επιτρέπει στα κράτη-μέλη να εμπλακούν, να συμμετάσχουν στη διαδικασία ε, της τη μεταφορά μια οδηγία. Είναι πάρα πολύ καινούργιο αυτό και αυτό ήταν πολύ ενδιαφέρον. Εάν δεν είχε υπάρξει αυτή η μέθοδος της αμοιβαίας αξιολόγησης, θα είχαμε παραμείνει νομίζω σε μια ανταλλαγή ε, μεταξύ γειτονικών χωρών που είναι συνηθισμένες να κάνουν τέτοιες ανταλλαγές μεταξύ τους διμερώς συνήθω. Ενώ έτσι μπορέσαμε όλοι να εκφραστούμε αυτή η διαδικασία αμοιφέας αξιολόγησης είναι κυρίως μια ε, ανταλλαγή εμπειριών για τη μεταφορά στο εθνικό δίκαιο. Όσον αφορά την οργάνωση της μεταφοράς αυτής στα κράτη-μέλη. Πώς οργανώθηκαν τα κράτη-μέλη για να μεταφέρουν ιδανικά την οδηγία αυτή. Στη Γαλλία αυτό έγινε σε επίπεδο δια υπουργικό, διπουργικό, σε κάθε υπουργείο που αφορά το από την οδηγία αυτή υπήρχε ένας υπεύθυνο και εξ αυτού έγινε και μία ανταλλαγή εμπειριών και απόψεων με άλλα κράτη-μέλη. Πολύ αποτελεσματική μέθοδος. Η ανταλλαγή εμπειριών όσον αφορά την ερμηνεία της οδηγίας για τις υπηρεσίες. Είχε τη Γαλλία η αμοιβή αυτή αξιολόγηση μας επέτρεψε σε περισσότερες ε, περιπτώσεις να επιβεβαιώσουμε τις επιλογές που είχαμε κάνει κατά τη μεταφορά αυτά της οδηγίας. Αυτή η διαδικασία είναι και μια δυνατότητα να υπάρχει μια καλύτερα ορατότητα των ε, τροποποιήσεων ε, των διαγραφών που έγιναν στην οδηγία αυτή και να εξτάσουμε επίσης τι ήταν δικαιολογημένο να γίνει και τι όχι. Το σύστημα αυτό συνενώνει όλα τα διάφορα σημεία και ε, αποτελεί ένα σύνολο πλουσίων ε, εμπειριών. Είναι δύσκολο όμως γιατί ε, είδαμε υπήρξαν δεκάδες χιλιάδων δελτία που συμπληρώθηκαν για το θέμα αυτό. Αυτό ήταν το πρώτο πρόβλημα ο τεράστιο αριθμός δηλαδή των δελτίων που είχαν συμπληρωθεί, Εκτό αυτού τα δελτία αυτά ήταν συμπληρωμένα στην εθνική γλώσσα του εκάστοτε κράτου μέλους. en euh, Χρειάστηκε λοιπόν να γίνει μια συνεδρίαση ολομέλειας για να γίνει κατανοητό αυτό το σύστημα. Εδώ και βέβαια μια βοήθεια για την μετάφραση των δελτίων αυτών στα αγγλικά τουλάχιστον και αυτό οπωσδήποτε επέτρεψε να εκμεταλλευτούμε αυτή τη βάση πληροφοριών έτσι είχαμε βέβαια πιο σύντομη περίοδο αμοιβαία αξιολόγηση, αλλά δεν μπόρεσαν να γίνουν άμεσε ανταλλαγέ μεταξύ των κρατών μελών απαραίτητο. Κατόπιν, όσον αφορά τα αποτελέσματα της αμοιβαίας ε, αξιολόγησης, η ανακοίνωση Κομισιόν έδειξε ότι υπήρχαν προβλήματα, το υπενθυμίσαμε αυτό, η Κομισιόν προτείνει επίσης κάποιες πρωτοβουλίες, κάποιες δράσεις. Παραδείγματο χάρη είναι έναν έλεγχο της ε, ε, πρακτική οδηγή. Θεωρώ λοιπόν ότι όλες αυτές οι δράσεις επέτρεψαν την διατήρηση διαλόγου μεταξύ των κρατών μελών αφενός και μεταξύ των κρατών μελών και της Επιτροπής Αφετέρου και αυτό είναι κάτι που πρέπει να το διατηρήσουμε και για το μέλλον μου φαίνεται. Ευχαριστώ πολύ. Πρόεδρος, εγώ σας ευχαριστώ για τις ε, για τον λεπτομερή τρόπο με τον οποίο μας παρουσιάσετε τα θέματα. Ερωτήσεις αργότερα. Τώρα κάποιο που ενεπλάκει στη διαδικασία, η κυρία Βίλ Σεμπαρκότσκα από την Πολωνία. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Εκπλήττω που μπορώ να ακούσω πολωνικά εδώ. Θα μιλήσω όμως αγγλικά, γιατί έχω παρουσιάσει, ε, προετοιμάσει την παρουσίασή μου στα αγγλικά. Και στα πολωνικά μου χρησιμοποιώ αγγλικές λέξεις. Ε, δεν είναι πολύ καλό αυτό και λυπούμε που δεν θα ε, χρησιμοποιήσω τη δυνατότητα να μιλήσω τη μητρική μου γλώσσα που μου προσφέρετε. Καταρχήν θέλω να σας πω ότι όλη αυτή η διαδικασία συζήτηση για την ε, οδηγία της υπηρεσία και η μεταφορά αυτή στο εθνικό δίκαιο και η αμοιβαία αξιολόγηση ήταν μια πάρα πολύ αξιόλογη εμπειρία. Πολλά μάθαμε και μάθαμε επίσης πώς οργανώνονται οι υπηρεσίες αυτές διαφορετικά και αντιμετωπίζονται διαφορετικά σε διάφορα κράτη-μέλη. Η αμοιβή αυτή αξιολόγηση ήταν για μας ένα πολύ ακριβό σύστημα και ένα πολύ χρονοβόρο σύστημα. Το λέω αυτό γιατί αναφέρεται και στην έκθεση. Και το συζητήσαμε μεταξύ μας, είδαμε πραγματικά πόσο χρόνο χρειαζόμασταν γι' αυτό. Οι εμπειρογνώμονες ε, εργάστηκαν σκληρά για να αναλύσουν πάρα πολλά στοιχεία, πάρα πολλές εκθέσεις και να συμμεριστούν αυτά τα αποτελέσματα με τις εθνικές διοικήσεις και με τα άλλα υπουργεία που αφορούσε αυτή τη διαδικασία. Εκτιμούμε ιδιαίτερα την βοήθεια της Κομισιόν και την αόρατη χείρα βοηθείας που μας έτεινε. Μπορούσαμε να μιλήσουμε ελεύθερα κατά τη διάρκεια της διαδικασίας αυτής και μάθαμε πολλά ημέν από τους δε. Για μας, αυτό ήταν το πιο αξιόλογο. Είμαστε στο ίδιο κλάστερ όπως η Γερμανία. που είναι ο κύριος μας ε, ε, γείτονας ε, εμπορικός εταίρος, η κυρία μας πηγή θα έλεγα. Και ήταν πολύ ενδιαφέρον να δούμε πόσο ο τομέας είναι οργανωμένος στην Γερμανία, να κατανοήσουμε έτσι τα προβλήματα και μας βοηθάει επίσης να δούμε ότι τα πράγματα δεν είναι τόσο εύκολα και τώρα καταλαβαίνουμε γιατί δεν είναι τόσο εύκολα. Αυτό είναι ένα πάρα πολύ θετικό στοιχείο της διαδικασίας που πρέπει να έχουμε κατά νου. Τώρα, η συνέχεια που πρόκειται να δοθεί, το πρώτο ερώτημα που αναφέρεται, είναι σημαντικό νομίζω να έχουμε κατά νου το εξή. Γνωρίζουμε πολλά ημέρια τους ΔΕ αλλά είναι και πάρα πολύ σημαντικό τι θα κάνει από εδώ και πέρα η Κομισιόν. Δηλαδή, ποια θα είναι η οικονομική αξιολόγηση της εφαρμογής της οδηγίας για τις υπηρεσίες. Αυτό κατά γνώμη μας είναι πάρα πολύ σημαντικό. Και αυτό είναι ένα βήμα που χρειαζόμαστε. Γιατί το να πούμε ότι αυτή όλη η διαδικασία που είναι τόσο πολύπλοκη, με τη, πολύπλοκη μεταφορά, της ε, μεγάλες προσπάθειας που έχουν καταβληθεί για την αμοιβαία αξιολόγηση. Θα πρέπει να καταμετρήσουμε το κόστος της διαδικασίας σε σχέση με την αξία, με το όφελος που απορρέει από αυτά. Ότι δηλαδή η αγορά θα μπορέσει να κινείται πιο ελεύθερα ε, πέρα από τα σύνορα. Εγώ στο Υπουργείο Οικονομικών είμαι υπεύθυνη για τα μέσα της ε, λειτουργίας αγορά, της εσωτερικής αγοράς. Δεν βλέπω πολλούς να κάνουν ε, πολλές κινήσεις προς την κατεύθυνση αυτή. Γιατί όμως, γιατί είναι τόσο καλά τα πράγματα ή γιατί δεν κινούνται πολύ διασυνοριακά. Η οδηγία αυτή ψηφίστηκε το 2006. Υπήρχαν τρία χρόνια διαθέσιμα για την μεταφορά στο εθνικό δίκαιο και τώρα έχει περάσει άλλος ένας χρόνος από τότε. Και η δική μου προσωπική εμπειρία δεν με έκανε να δω να υπάρχει μια πραγματική κίνηση στην αγορά προσφοράς υπηρεσιών και γιατί, γιατί αυτό με ενδιαφέρει. πάλι σας ευχαριστώ για αυτές τις παρατηρήσεις. Θα δούμε στο τελευταίο σημείο μερικές από αυτές. Τώρα, επόμενη Επόμενη ομιλήτρια είναι η κυρία Στραντμπάκε από την Σουηδία την καλά. Σωρίζουμε εδώ μετά από ένα μακρύ ταξίδι. Σας δίνω το λόγο για πέντε λεπτά. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ την Επιτροπή ε, για την πρόσκληση. Χαίρομαι που είμαι εδώ για να μιλήσουμε για την αμοιβαία αξιολόγηση. Ήμουνα στην προηγούμενη μελέτη ως σημείο εκκίνησης για αυτήν ε, την ε, συζήτηση ε, μπορώ να πω ότι υποστηρίζουμε τη μέθοδο. Αυτή η μέθοδος συνέβαλε σε εφαρμογή διαφανέστερη και αποτελεσματικότερη Είχαμε μια μέθοδο πριν από το 2009. Δεν ξέρω αν η μέθοδος αμοιβαίας αξιολόγησης μπορεί να δώσει χρήσιμα αποτελέσματα. Ε, βεβαίως χρειάστηκε να κάνουμε μια επιλογή ανάμεσα στα κράτη-μέλη και να αξιολογήσουμε πολλά στοιχεία, 35.000 ε, και είχαμε ακόμα και το θέμα των κοινοτικών ε, γλωσσών, αλλά ευτυχώς ε, μπορεί κανείς να αλλάξει γνώμη και η διαδικασία αυτή δεν μας τρομάζει τόσο όσο προηγουμένως. Διαπιστώσαμε ότι η διαδικασία αυτή ήταν χρήσιμη και μας επέτρεψε να έχουμε απτά αποτελέσματα. Όπως ανέφερε και η Κομισιό, η αμοιβαία αξιολόγηση από την δική μας άποψη είχε επιπτώσεις πάνω στην ενιαία αγορά ε, στην Σουηδία όταν ζητήσαμε από τις εθνικές δικήσεις να αξιολογήσουν τα κριτήρια από την άποψη της ενιαίας αγοράς. Για μας ε, η μέθοδος αυτή επέτρεψε να ε, δημιουργήσουμε ένα διάλογο μεταξύ των κρατών μελών, έφερε την διαφάνεια και μπορέσαμε να αναδείξουμε τις βέλτιστες πρακτικές. Όσο προς τα αποτελέσματα που πετύχαμε, χαιρετίζουμε την ακοίνωση Κομισιό που δημοσιεύθηκε στην αρχή του έτους και επέτρεψε τη συζήτηση μεταξύ της ομάδας εμπειρογνωμόνων που τόνισαν ποια είναι τα σημεία που πρέπει να επισύρουν περισσότερο την προσοχή δόθηκε σημασία στις δραστηριότητες υπηρεσιών που περιορίζονται σε μερικούς φορείς χωρίς κανέναν ιδιαίτερο εμφανή λόγο πολιτικής. Άλλο σημαντικό σημείο της αμοιβαία αξιολόγησης είναι η ε, χρησιμοποίηση κοινή οικονομικής βάσης που ε, εφαρμόζεται πολύ από τα κράτη-μέλη παρά την απαγόρευση. Θα πρέπει να εξασφαλίσουμε την ε, παρακολούθηση της εφαρμογής ε, της οδηγίας για τις υπηρεσίες. Τα αποτελέσματα της αξιολόγησης επέτρεψαν να δούμε ότι το θέμα αυτό είναι επίγον και χαιρετίζουμε τα συμπεράσματα του Συμβουλίου του Μαρτίου που ζητά μεγαλύτερη προσοχή για τον τομέα των υπηρεσιών. Πρέπει οπωσδήποτε να διατηρήσουμε την όθηση την οποία συσσωρεύσαμε για αυτήν την οδηγία και χαίρομαι που η Επιτροπή έχει ασχοληθεί με το θέμα αυτό. Ευχαριστώ, ευχαριστώ για τα σημαντικά αυτά σημεία. Θα επανέλθουμε σε το θέμα αυτό των ορισμένων επαγγελμάτων, ορισμένων τομέων. Να δούμε αν θα έχουμε μια αλληλεπίδραση μεταξύ σας. Και τέλος, Χαιρετίζω ε, την Ατελή Ζουάν που δεν είχε να αντιμετωπίσει τον νέφος της τέφρα σήμερα. Ήρθε ίσως με λεωφορείο, δεν ξέρω. Ήρθε από το Παρίσι. Θα ήθελα να ευχαριστήσω την Επιτροπή αυτή της ενιαίας αγοράς της και των καταναλωτών για την πρόσκληση. Θέλουμε εδώ ένα feedback για να δούμε τι γίνεται με τις εθνικές δικήσεις. Θα ήθελα πρώτα απ' όλα να τονίσω ότι η περιοχή δεν έχει οθετήσει επίσημη ε, θέση για την αξιολόγηση την αμοιβαία. Γι' αυτό μιλάω προσωπικά και θα ήθελα να πω με ποιον τρόπο στο Βέλγιο που είναι ομοσπονδιακό κράτος αντιμετωπίσαμε το θέμα αυτό της μεταφοράς διότι η διαδικασία αμοιβαία αξιολόγησης ήταν μια παράταση των δομών που είχαν θεσπιστεί για την μεταφορά στο εθνικό δίκαιο, για την μεταφορά το, η κάθε οντότητα είχε μια αυτονομία στην μέθοδο μεταφοράς και είχαμε ένα συντονισμό με μια πλατφόρμα στο Ομοσπονδιακό Υπουργείο Οικονομίας. Δεν υπήρχε τυπική σχέση ανάμεσα στις διάφορες οντότητες για να εξασφαλιστεί η μεταφορά και η διαδικασία της αμοιβαία αξιολόγησης. Σχετικά με την διαδικασία αυτή ε, δεν ήταν δυνατό να είμαστε οκτώ γύρω από το τραπέζι. Ήμασταν απλώς τρεις περιφέρειες ε, του Βελγίου και το επίπεδο το ομοσπονδιακό εκπροσώπησε τις αρχές μας. Όσον αφορά το κλάστερ, ήμασταν με τη Γαλλία, το Λουξεμβούργο, το Λίχτενστάιν και τις ε, κάτω χώρες. Ήμασταν από τις λίγες χώρες που είχαμε επίσημο εκπρόσωπο μια μικρή διευκρίνηση για να εξασφαλίσουμε την διαδικασία μεταφοράς και την διαδικασία αμοιβαία αξιολόγησης, δημιουργήθηκε μια έκτακτη ad hoc μονάδα στην περιφέρεια των, της πρωτεύουσας Βρυξέλλες, Καπιτάλ Καπιτάλ, για τον συντονισμό της αμοιβαία αξιολόγησης. χρειάστηκε να αναπτύξουμε δίκτυα, να συγκεντρώσουμε την πληροφορία που ήταν μια εργασία πλήρους απασχόλησης για την μεταφορά και την αμοιβαία αξιολόγηση. Νομίζω ότι είναι σημαντικό να τονίσουμε ότι για να έχουμε αντίκτυπο συγκεκριμένο ότι όσον αφορά την διαδικασία αμοιβαία αξιολόγησης μπορούμε να πούμε για την περιφέρεια ότι η εμπειρία ήταν γενικά θετική. Πρέπει επίσης να πούμε ότι ως προς την παρακολούθηση της ευρωπαϊκής οικονομικής πολιτικής δεν υπήρχε πραγματογνωμοσύνη εσωτερική στο επίπεδο της περιφέρειάς μας και δεν ξέρω πώς γίνεται σε, άλλες, σε άλλα ομόσπονδα κράτη ε, και σε ομοσπονδιακό επίπεδο Το σημείο αυτό είναι σημαντικό, η μεταφορά και η αμοιβαία αξιολόγηση υπήρξαν ε, κάτι το καλό για να δημιουργηθεί ένα δίκτυο, να διαδοθούν ιδέες μέσα στη δίκηση και μεταξύ των συναδέλφων μου. Θα ήθελα να πω ότι ο φόρτος εργασίας ήταν σημαντικός, είναι ένα αντικειμενικό στοιχείο. Η παιδαγωγική εργασία που πρέπει να κάνουμε εσωτερικά ως υπάλληλοι απέναντι στους συναδέλφους και αυτό δείχνει ότι η αμοιβαία αξιολόγηση είναι μια καλή διαδικασία ε, διότι και εμείς έτσι μπαίνουμε σε μια φάση μαθητείας και συνεργασίας με τους Ευρωπαίους συναδέλφους. Κάτι το θετικό. Είχαμε δυσκολίες σε γλωσσικό επίπεδο βεβαίως, εφόσον όλοι οι υπάλληλοι ε, όλοι δεν μπορούν να εργαστούν στα αγγλικά και να συντάσσουν εκθέσεις στα αγγλικά. Στο επίπεδο των αποτελεσμάτων πρέπει να δούμε επίσης και τις περιφερειακές αρμοδιότητες και τι μέσα υπάρχουν ε, στην, στον περιβαλλοντικό τομέα, στην οικοδομή, στον τουρισμό, την ρύθμιση που υπάρχει στα ταξιδιωτικά γραφεία και τα επαγγέλματα που ήταν στο επίκεντρο των συζητήσεων μεταξύ συναδέλφων. Αυτά νομίζω ότι πρέπει να πούμε ότι για μας δεν ήταν πάντοτε προφανές να, ότι έπρεπε να επικοινωνούμε ε, για ε, κανονισμούς που ήταν ε, αντικείμενα συζητήσεων σε περιφερειακό κοινοβούλιο σε επίπεδο, ή σε επίπεδο ομοσπονδιακό. Έτσι ήταν και η κατάσταση και στην περιφερειά μας και σε άλλα κράτη-μέλη και αυτό καθιστούσε δύσκολες τις ανταλλαγές, ενδιαφέρουσες αλλά δύσκολες, αλλά και όπως λέχθηκε από τους εμπειρογνώμονες που ασχολήθηκαν με την συνολική μελέτη για την διαδικασία, είναι αληθές ότι μετά την διαδικασία αμοιβαία αξιολόγησης μπορεί κανείς να σκεφτεί ότι πρέπει να αλλάξει προσανατολισμό, να επιφέρει τροποποίησης, αλλά είναι τότε πολύ αργά. Και ίσως θα πρέπει σε 4 ή 5 χρόνια ε, να τροποποιηθούν ορισμένα πράγματα, αλλά δεν μπορούμε τώρα να τροποποιήσουμε κάτι που μόλις τροποποιήθηκε. Πρέπει όμως να διατηρήσουμε τη γνώμη και την, την γνώση και την πραγματογνωμοσύνη. Δεν είναι προφανές. Δεν ε, μπορεί να γίνει επίσης και η διαδικασία αμοιβαίας αξιολόγηση στην περίοδο της ε, μεταφοράς. Εγώ αυτό που συγκρατώ τελικά είναι ότι λόγω αυτής της ε, μεταφράστης της οδηγίας για τις υπηρεσίες και τις διαδικασίες αμοιβές αξιολόγηση υπάρχει στη δική μας ε, περιφέρεια Μπρουσέλ Καπιτάλ μια προστιθέμενη αξία και σταθεροποιείται ο συντονισμός ο οικονομικός μέσα στην περιφέρεια και έχουμε προστιθέμενη αξία σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ που μοιραστήκατε αυτές τις ιδέες σας. Βλέπουμε κοινά, βλέπουμε διαφορές και είναι πολύ ενδιαφέρον και για μας. Ερωτήσεις από συναδέλφους και βεβαίως εάν και ο καθηγητής Μπερζέ ε, έχει κάποιες ερωτήσεις ε, φυσικά ή κάποια σχόλια φυσικά. Θα δώσω το λόγο πρώτα απ' όλα στην κυρία Γκέμπχαρτ γιατί μην ξεχνάμε ότι είναι και η συγγήτρια. Να μοιραστεί σκέψεις και σχόλια μαζί μας. Άκουσα καταρχήν με πάρα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Θα ήθελα να πάω δύο-τρία βήματα προς τα πίσω και να σας υπενθυμίσω ότι ήταν πολύ σκεπτικό το κοινοβούλιο όσον αφορά αυτό το σύστημα της αμοιβαίας αξιολόγησης. Ε, το είχε προτείνει η Κομισιόν, το, το Κοινοβούλιο το διάγραψε και τα κρατη το επανέφεραν. Αυτό είναι το ιστορικό, τι θέλω να σας το υπενθυμίσω. Ένας από τους λόγους για τους οποίους είμαστε κάπως επιφυλακτικοί ακούστηκε λιγάκι από τις διάφορες εκθέσεις. Το κόστος, η γραφειοκρατία και η εργασία που απαιτεί αυτό και κατά πόσον όλα αυτά πραγματικά είναι χρήσιμα, αν τα δούμε σε σχέση κόσοφελίας, ή αν θα ήταν κατάλληλα κάποια άλλα μέσα. Τώρα ακούω πολύ θετικά σχόλια για τις εμπειρίες αυτές και αν υπάρχει κάτι τέτοιο, το αποτέλεσμα είναι πάρα πολύ θετικό προφανώς. Και θα ήθελα να επανέλθω σε αυτό που είπε η κυρία Ζουά μόλις τώρα. Τι θα γίνει από εδώ και πέρα, σε 2, 3, 4, 5 χρόνια. Είπατε ότι ορισμένα άτομα έχουν κάνει αυτές τις εμπειρίες. Έχουμε την εμπειρία, ξέρουμε πώς θα μπορούσαν να προχωρήσουν τα πράγματα. Τι θα γίνει όμως σε πέντε χρόνια αν αυτά τα άτομα δεν έχουν αυτές τις θέσεις πια. Ποιος θα, θα θυμηθεί αυτά όλα. Ποιος θα θυμάται τι είχε γίνει. είναι μόνιμες οι εντυπώσεις ή παραμένουν μονάχα εφόσον εξακολουθούν να υπάρχουν τα άτομα που έκαναν αυτές τις εμπειρίες. Από όσο κατάλαβα εγώ διαβάζω στα έγγραφα, είδα σε ορισμένα κράτη-μέλη ήταν τα Υπουργεία υπεύθυνα, αλλά θα μείνει αυτή η μνήμη αν θέλετε, αλλά υπάρχουν και άλλα κρατημέλη που προσέλαβαν κάποιου εξωτερικούς συνεργάτες για να κάνουν την εργασία αυτή. Και θα ήθελα πραγματικά να ξέρω εσείς πώς το αξιολογείτε. Τι είναι το καλύτερο. Το δεύτερο ερώτημα, γιατί κοίταξα τα πράγματα εδώ στα γλίγορα και αυτά εδώ πέρα που μας είχαν αποστείλει. Και ο κύριος Όμπερντορφ μας έστειλε το έγγραφό του στα γερμανικά. Για μένα αυτό είναι πολύ πρακτικό. Και διαβάζω ακριβώς ε, το αντίθετο αυτών που άκουσα μέχρι στιγμής. Είναι πραγματικά πολύ λυπηρό που δεν είναι παρόν ο κ. Γιατί θα σας ε, παραθέσω μια πρόταση, πρώτη παράγραφο. Κατά τη διάρκεια της εφαρμογής ε, της ε, οδηγίας για τις υπηρεσίες υπάρχει και το σύστημα της αμοιβαίας αξιολόγησης, το οποίο οι περισσότεροι που συμμετείχαν σε αυτό θεώρησαν ότι είναι υπερβολικά γραφειοκρατικό και αναποτελεσματικό. Ακριβώς το αντίθετο δηλαδή αυτό που άκουσα. Εμένα θα με ενδιαφέρε πώς είναι δυνατόν να είναι τόσο διαφορετικές οι εμπειρίες από το σύστημα αυτό της αμοιβαίας αξιολόγησης. Και εδώ προσθέτω και μία άλλη ερώτηση προς όλους τους εμπειρογνώμενες. Κάτι που θα πει και ω Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Μέσα στα πλαίσια της ε, αξιολόγησης και του screening. Ότι δεν θα πρέπει να εξαρτώμεθα μόνο από το πολιτικό επίπεδο, αλλά σε συνεργασία με τους άμεσα ενδιαφερόμενους. Δηλαδή μαζί με εκείνους που προσφέρουν τις υπηρεσίες, κατά πόσον έχουν συμπεριληφθεί οι εμπειρίες τους, αλλά και οι εμπειρίες των καταναλωτών και των εργαζομένων. Το πρώτο που θέλαμε να πετύχουμε να υπάρχει ελευθερία της προσφοράς των υπηρεσιών, να υπάρχει ελεύθερη κυκλοφορία, αλλά να υπάρχουν και κάποιοι απαραίτητοι κανόνες που να τηρούνται πράγματι. Δεν άκουσα πολλά από αυτού και θα ήταν καλό να μου δίνατε κάποιες συμπληρωματικές πληροφορίες. Θα επανέλθουμε και στους εμπειρογνώμονες και στην εκπρόσωπο της Κομισιόν σε λίγο. Η Ευχαριστώ πολύ. Κύριε Πρόεδρε, θα ήθελα πρώτα απ' όλα να ευχαριστήσω όλους τους ε, εμπειρογνώμονες για αυτή την ενδιαφέρουσα εμπειρία ε, που ε, βασίζεται στις δικές τους εμπειρίες ε, όσον αφορά την αμοιβαία αξιολόγηση. Έχω την εντύπωση Για, έχω την εντύπωση ότι εδώ ακούσαμε πολλές βέλτιστες πρακτικές. Ήταν μια άσκηση πολύ μυητική κατά κάποιο τρόπο στην όλη διαδικασία και είμαστε πλέον σε θέση, νομίζω, να βελτιώσουμε και την ομολογία, δηλαδή να εισαγάγουμε πιο έξυπνη ε, νομοθεσία η οποία με καλύτερο τρόπο θα προσαρμόζεται στις ανάγκες ε, των οικονομικών ε, φορέων. Έχω πάντως ακόμα κάποια ερωτήματα για τους πανελίστες και τους εμπειρογνώμονες. Ερώτηση πρώτη. Η διαδικασία αμοιβαία αξιολόγηση έλαβε χώρα σύμφωνα με, την, με τα όσα προβλέπονται στην οδηγία. Αληθεύει ότι το μοντέλο αυτό τελικά μείωσε την ε, ε, μεταφορά της οδηγίας θα ήταν καλύτερα να είχε ξεκινήσει νωρίτερα η διαδικασία έτσι ώστε τελικά ε, να είναι καλύτερος ο αντίκτυπος όλων αυτών των προνοιών ε, προς όφελος, τα, των κρατών μελών. Επίσης, τα κράτη-μέλη που είναι παρόντα εδώ και έχουν τέτοια εμπειρία να μου πούν ποια είναι η γνώμη σας όσον αφορά την σύσταση των κλάστερς. Πιστεύετε ότι θα είχε δουλέψει καλύτερα το σύστημα των κλάστερς εάν η σύνθεση των κλάστερς αυτών ήταν διαφορετική. Τα κράτη-μέλη είχαν επιλογή όσον αφορά τα clusters. Τέλος, μια ερώτηση προς την εκπρόσωπο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή προτίθεται να χρησιμοποιήσει τα αποτελέσματα αυτής της διαδικασίας αμοιβαίας αξιολόγησης. Κατανοώ ότι η όλη διαδικασία βοήθησε την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να καταλάβει, να κατανοήσει καλύτερα το περιεχόμενο της αξιολόγησης. Αλλά ε, έχει στοιχεία η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ε, μετά από αυτές τις αμοιβές αξιολογήσεις ότι εφαρμόστηκε καλά η οδηγία ότι οι διαδικασίες, ε, οι, τον, επίσης οι διαδικασίες ανάμεσα στα κράτη-μέλη τα οποία δεν εφήρμοσαν την οδηγία αυτή θα είναι διαφορετικές. Για μία ακόμα φορά σας ευχαριστώ. Ευχαριστώ τους εμπειρογνώμονες που ήρθαν και έκαναν τόσο ενδιαφέρουσες παρουσιάσεις. Ευχαριστώ πολύ. Θα ήθελα και εγώ να κάνω κάποια σχόλια και ως σκιώδη συγητή της εκθέσεως Γκέπχαρτ για την οδηγία για τις υπηρεσίες αλλά και γιατί άκουσα με ενδιαφέρον και θέλω να κάνω κάποιες προτάσεις. Νομίζω ένα από τα ενδιαφέροντα ε, σημεία ε, είναι το ότι έχουμε δύο ε, επίσης από τους εμπλεκόμενους φορείς παρόντες εδώ, αλλά νομίζω κάτι που δεν πρέπει να ξεχνάμε στις διαδικασίες ε, αξιολόγησης είναι το να ακούμε την άποψη των συμμετεχόντων. Η διαφάνεια της διαδικασίας είναι πολύ σημαντική γιατί νομίζω ότι η διαδικασία ήταν μάλλον κρατική, διακυβερνητική. Δημιουργήσατε όμως δίκτυα, σχέσεις μεταξύ σα, μιλούσατε ο ένας με τον άλλον και ε, ε, αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Σε μερικές περιπτώσεις ε, κάποιοι από τους εμπλεκόμενους είχαν και άποψη σχετικά με το πώς θα δημιουργεί το, η ομάδα. Αλλά νομίζω ότι και το κεντρικό ερώτημα είναι, και αυτό είναι αντίθετο προς αυτό που είπε η κυρία Χάσλικ προηγουμένως, ε, ίσως ξεκίνησε πολύ ε, νωρίς η διαδικασία γιατί δεν είχαν προβλήματα οι εμπλεκόμενοι μέχρι να αρχίσει να εφαρμόζεται η οδηγία. Φαίνεται ότι ε, υπήρξε μία απογοητευτική τροπή τελικά ε, όσον αφορά την ίδια την οδηγία και ε, το τι έγινε μετά την ε, μεταφορά της οδηγίας. Ενδεχομένως το πρόβλημα ήταν και ψυχολογικό λίγο, αλλά πάντως νομίζω ότι το, το θέμα της διαφάνειας, το θέμα του, του κατά πόσον αναμίχθηκαν ή όχι οι εμπλεκόμενοι φορείς, αυτά είναι τα κυρία ζητήματα. Και επίσης ε, πολύ σημαντικό είναι το ζήτημα του ποιοι συμμετείχαν στην ε, διαδικασία. Σε άλλες χώρες, ε, δηλαδή σε κάθε χώρα διέφεραν οι συμμετέχοντες. Νομίζω ότι είναι πάρα πολύ ενδιαφέρον να έχουμε και την άποψη των λοιπόν εμπλεκομένων. Έχουμε άλλες ερωτήσεις. Ο κύριος Βάμπ, θέλετε να ρωτήσετε κάτι? Ναι, θέλει ο κύριος Βάμπ, παρακαλώ. Μία τελευταία ερώτηση και μετά θα απαντήσουν οι εμπειρογνώμονες. Καταρχήν, ε, ζητώ συγγνώμη που τηλεφωνούσα μόλις τώρα, Πρόεδρε, αλλά ξέρετε τι γίνεται κανένα φορά. Ε, θα ήθελα να αναφερθώ σε αυτό που έγραψε ο κύριος Σόπερντορφ ε, στο κείμενό του, το ανέφερε και η κυρία Γκέπερτ. Αν το καταλαβαίνω σωστά, η δική του νομοδότηση αναρωτιέται κατά πόσο η διαδικασία αυτή μπορεί να χρησιμοποιηθεί ευρέως. Η απάντηση είναι όχι, γιατί βέβαια δεσμεύονται πάρα πολλοί πόροι και ανθρώπινοι πόροι και δεν είναι πάντα δυνατό. Αλλά θα επανέλθω σε αυτό που είπε η εκπρόσωπο τη Πολωνία. Νομίζω ότι η οδηγία προσφορά υπηρεσιών δεν ήταν πολύ απλή και συναισθηματικά. Και αυτό που λέτε ότι η κατανόηση για τη δυσκολία εφαρμογή τη οδηγία από την άλλη πλευρά των συνόρων προωθείται θετικά με την ε, διαδικασία αυτή της αμοιβαία αξιολόγησης. Άρα ήδη έχουμε ένα θετικό αποτέλεσμα της αμοιβαία αξιολόγησης. Και αυτό θέλω να ρωτήσω τη συνάδελφο από την Πολωνία κατά πόσο θεωρεί ότι αυτή η διαδικασία γενικά είχε τον απαραίτητο αντίκτυπο στην κοινή γνώμη ότι ούτως ώστε όχι μόνο όπως ανέφερε και η Γκέπα οι αρμόδιοι υπάλληλοι έχουν καταλάβει περί τίνος πρόκειται, αλλά κατά πόσον το ευρύ κοινό έχει επίσης καταλάβει τα πράγματα καλύτερα. Okay, Ενδεχομένως να ακούσουμε κάποιες απαντήσεις από τους εμπειρογνώμονες ε, ανάποδα να ξεκινήσουμε και η εκπρόσωπος της Κομισιόν να ε, ξεκινήσει την επόμενη, το επόμενο κομμάτι. Ίσως καλό θα ήταν να ακούσουμε από τον καθηγητή ε, Μπερζέ και ή και από τον κύριο Πλάτ ορισμένα πράγματα σε σχέση με αυτά που ακούστηκαν η κυρία Μασάρ και θα συνεχίσουμε με τις υπόλοιπες ομιλήτριες. Ε, Καθηγητά Βεζέ, παρακαλώ. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Ναι, εγώ, εμείς έχουμε κατανέμει λίγο τις ε, ε απαντήσεις ε, σε σχέση με την ερώτηση κυρίας Γκέμπχαρτ. και σε σχέση και με αυτά που είπε η εκπρόσωπος του προγράμματος από την περιφέρεια Βρυξελών. Νομίζω ότι στην ε, οδηγία για τις υπηρεσίες η διαδικασία αφορά μονάχα ε, τα ορισμένα στοιχεία τα οποία βρίσκονται πάντα στο στόχαστρο ε, της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και της Ένωσης γενικότερα. Είτε οι διαδικασίες αυτές ε, μεταφέρουν απλώς ε, τα, την έκβαση της ομολογίας και το περιεχόμενο των ίδιων των συνθήκων ε, και που εξετάζονται με τον ένα ή τον άλλο τρόπο, δηλαδή είτε από νομικής απόψεως είτε από νομοθετικής απόψεως από τα ίδια τα θεσμικά όργανα, είτε στη, στην, στα πλαίσια της πολυτομιακότητας Εκεί ξέρουμε ότι θα πρέπει να ενισχυθούν ε, τα clusters, ε, θα πρέπει να ενισχυθεί η ε, περαιτέρω προσέγγιση μεταξύ των τομέων και να αποφύγουμε οποιαδήποτε απομόνωση. Αλλά βεβαίως είναι η υπηρεσία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής που θα πρέπει να προσπαθήσουν έτσι ώστε οι εμπλεκόμενοι φορείς, έτσι ώστε μάλλον να έρθουν πιο κοντά στους εμπλεκόμενους φορείς, έτσι ώστε ε, να κάνει η Κομισιόν καινούριε προτάσεις και για την επιμήκυνση της οδηγίας ή προς κάποια άλλη κατεύθυνση. Επομένως, το μετά βρίσκεται μεταξύ των χειρών της Ευρωπαϊκής Επιτροπής ή γενικότερα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αυτό μου φαίνεται προφανές. Δεύτερο ερώτημα στο οποίο θα απαντήσω τη Κυρία Χάνσλικ. Δηλαδή Μήπως θα έπρεπε να είχε ξεκινήσει η διαδικασία με βάση αξιολόγησης όχι μετά την θεωρητική τουλάχιστον μεταφορά της οδηγίας αλλά πριν. Η πραγματικότητα κατέδειξε ότι ωραία ανακατεύτηκαν όλα αυτά. Υπήρχαν κάποιοι οι οποίοι καθυστέρησαν, υπήρχαν χώρες οι οποίες προχώρησαν πολύ γρήγορα, άλλες προχώρησαν λιγότερο γρήγορα σε σχέση με άλλες ε, και επομένως δεν ε, ξεκίνησαν και ολοκληρώθηκαν όλες οι διαδικασίες μαζί και την ίδια χρονική στιγμή ε, υπήρχαν χώρες οι οποίες ε, εκμεταλλεύτηκαν ας πούμε την εμπειρία άλλων χωρών που προηγουμένως ε, είχαν ασχοληθεί με τα θέματα αυτά. Επομένως, λόγω ακριβώς του ότι δεν σεβάστηκαν τα κράτη-μέλη τις χρονικές διαδικασίες, υπήρξε μία ανάμιξη και μία επικάλυψη. Ε, οι εμπλεκόμενοι ενδεχομένω θα μπορούσαν να πούνε περισσότερα πράγματα, αλλά νομίζω ότι τρει είναι οι ερωτήσει και μάλλον συγκεκριμένε. Ε, ε, εκεί υπάρχουν ζητήματα, όχι στη γενικότερη ή στη συνολική μεταφορά της οδηγίας. Ε, βεβαίως, μπορούν να υπάρξουν, βεβαίως μπορεί να υπάρξουν ανταλλαγές, αλλά δεν ήταν ε, η αρχική φιλοδοξία του προγράμματος. Ε, το ζήτημα, προγράμματος, το ζήτημα είναι τι θα κάνουμε στο μέλλον, τι θα, γίνει, τι θα κάνουμε στο μέλλον βάσει της εμπειρίας που είχαμε μέχρι τώρα. Όσον αφορά την ερώτηση για την υλοποίηση της διαδικασίας, νομίζω ότι αυτό θα το συζητήσουμε στο δεύτερο σκέλος. Ευχαριστώ. Χωρίς μικρόφωνο. Α, ο κύριος Πλάτ. Σε σχέση με τα ερωτήματα που αφορούν την διαφάνεια, βεβαίως η διαδικασία αμοιβαίας αξιολόγησης δεν παρουσίαζε μεγάλο βαθμό ε, ε, διαφάνειας. Περιμέναμε ε, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να κοινοποιήσει τα αποτελέσματά της για να δούμε. Υπάρχουν λοιπόν δισταγμοί όσον αφορά την διαφάνεια. Τώρα, ε, σε σχέση με τα clusters οι διαδικασίες και οι συζητήσεις είτε έγιναν παρουσία της Κομισιόν είτε άνευ ήταν ε, ε, σοβαρές συζητήσεις με, με ανταλλαγή απόψεων οι ανταλλαγές ήταν αρκετά ανοιχτές, αρκετά ειλικρινείς ε, και νομίζω ότι θα μπορούσαν να είναι πολύ περισσότερο ε, ειλικρινής και ανοιχτή, θα μπορούσε να είχε πνεύσει ένας αέρας πιο ευρωπαϊκός, πράγμα που δεν ε, διαπιστώσαμε. Το ζήτημα είναι ότι θα έπρεπε να είμαστε σε θέση ανα πάσα στιγμή να παρακολουθούμε την διαδικασία, ε, που βρίσκεται η διαδικασία, σε ποιο στάδιο βρίσκονται οι συζητήσεις. Ε, ε, Τώρα είναι γεγονός ότι αρκετές χώρες απήντησαν στη διαβούλευση που ξεκίνησε η Κομισιόν, αλλά πρέπει να πούμε ότι οι ενδιαφερόμενοι έχουν διαφορετικό βαθμό αντιμετώπισης της διαφάνειας ή όχι. Δηλαδή δεν επικρίθηκε και γενικότερα η έλλειψη διαφάνειας. Δηλαδή δεν επέκριναν την διαδικασία αμοιβές αξιολόγησης για έλλειψη διαφάνειας, ενώ ε, υπήρξαν και οργανώσεις οι οποίες ήταν πιο εθνικές, ε, οι οποίες ε, δεν είχαν καθόλου τη δυνατότητα να εκφραστούν. Αυτές όντως επέκριναν τη διαδικασία αξιολόγησης για έλλειψη διαφάνειας. Ε, το, το σημαντικό ήταν να, ότι υπήρχαν οργανώσεις οι οποίες μπορούσαν να παρακολουθήσουν χωρίς να είναι παρούσες στις διαδικασίες, να γνωρίζουν την έκβαση των συζητήσεων, επίσης ο βαθμός απορρίτου των κρατών μελών ε, υπάρχουν πράγματα τα οποία δεν αποκαλύπτονται ε, στη διάρκεια αυτών των ανταλλαγών. Όσον αφορά την, ε, τις Βρυξέλλες, η διοίκηση είδε πάντα αυτή τη διαδικασία αμοιβές αξιολόγησης σαν μια διακυβερνητική διακρατική εργασία και επομένως υπήρχε διαφάνεια ε, ως ήθιστε στις δημοκρατικές ε, διαδικασίες, δηλαδή διαβούλευση με το Κοινοβούλιο, ε, με Υπουργεία κτλ. Δεν μας απασχόλησε πολύ περισσότερο όλο αυτό το θέμα, δηλαδή δεν θεωρήσαμε ότι θα έπρεπε να βρούμε κάποια ειδική διαδικασία. Όσον αφορά τη σύνθεση των κλάστερς, Πρώτα κάναμε εργασία σε κλάστερς και μετά στην ε, Ολομέλεια. Βεβαίως στα κλάστερς δουλεύουμε ε, σε άμεση συνεργασία με τις ε, εμπλεκόμενες χώρες. Γίνεται η διασυνοριακή συνεργασία πιο αποτελεσματική. Γνωρίζονται οι υπηρεσίες. Εμείς στο δικό μας κλάστερ πήγαμε αρκετά καλά. Μια παρατήρηση που κάναμε σαν Βέλγιο η παρουσία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στη διάρκεια της εργασίας σε κλάστερ, αλλά νομίζω ότι εδώ το πρόβλημα αφορά το Βέλγιο και την ε, ικανότητα της χώρας να μεταφέρει την ε, οδηγία. Εκεί είχαμε κάποια προβλήματα ε, και ψέξαμε την Επιτροπή γιατί δεν ήταν αρκετά παρούσα στην φάση κλάστερ θεωρήσαμε ότι μερικές φορές μάλιστα ε, η συμμετοχή της Ευρωπαϊκής Επιτροπής άλλαζε κατά κάποιο τρόπο την ε, ε, δυναμική του κλάστερ γιατί όποτε ήταν παρούσα έδινε παρόλα αυτά την ερμηνεία της όσον αφορά τις διάφορες φάσεις και τις διάφορες αποφάσεις ε, ενώ κατά την άποψή μου δεν θα πρέπει οπωσδήποτε να γίνεται αυτό στα κλάστερ ε, γιατί στην Ολομέλεια προβλέπεται η θέση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής αυτή ήταν μια δικιά μας άποψη σχετικά με το περιεχόμενο των συζητήσεων στα κλάστερς. όλες οι διαδικασίες, διαργασίες, ε, προϋποθέσεις, όροι που ε, μεταδίδονται στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή μέσω του IPM, κάποια ειδικά στοιχεία ε, ας πούμε για τη δικιά μας περιφέρεια, ή υπηρεσίες προς τις επιχειρήσεις κυρίως. Επίσης στον τομέα του περιβάλλοντος. Και νομίζω ότι κατά την άποψή μου πολύ σύντομα, πολύ γρήγορα, ε, τα νομικά ζητήματα τα αφήσαμε λίγο πίσω. Τα αφήσαμε λίγο παραπέρα λοιπόν, τα παραβλέψαμε όλα αυτά τα νομικά ζητήματα είναι γεγονός ότι μερικές φορές υπήρχε σύγχυση ε, για το τι κάνουμε, δηλαδή μεταφορά, αποτελεσματικότητα, τι θα κάνουμε, τι πρέπει να περιλαμβάνουν οι συζητήσεις μας. Όσον αφορά το ερώτημα τι μέλη γενέστε, τι θα γίνει μετά. Νομίζω ότι αυτό που είναι σημαντικό είναι να αναπτυχθεί ε, μια πραγματογνωμοσύνη η οποία θα σταθεροποιηθεί και η οποία θα μπορέσει να βοηθήσει πραγματικά τους εμπλεκόμενους φορείς. Ευχαριστώ. Ας, συνεχίσουμε σε Το πρώτο μου όνομα ε, Will ε, είναι πολύ πιο εύκολο. Το άλλο είναι αρκετά περίπλοκο. Θα ήθελα να σκεφτούμε λίγο για το θέμα των ενδιαφερομένων ε, μερών και της διαφάνειας ε, ε, στην αμοιβαία αξιολόγηση. Θα μπορούσαμε να θεωρήσουμε την συζήτηση ως ότι μπορούμε να έχουμε την αμοιβαία αξιολόγηση όταν συναντούμε ε, τις εθνικές δικήσεις των άλλων κρατών μελών, όταν η διαδικασία συνεχίζεται, διότι έτσι μαθαίνουμε ημένα από τους δε, βλέπουμε το πόσο περίπλοκο είναι αυτό από νομικής απόψεως και μετά μπορούμε να ε, χρησιμοποιήσουμε τις βέλτιστες ε, πρακτικές, να δούμε μερικές ομοιότητες και νομίζω, κατά τη γνώμη μου, θα μπορούσαμε να επηρεάσουμε όλη την διαδικασία ε, προς ε, μία ε, θετική κατεύθυνση όσον αφορά τη μεταφορά. Όταν γίνεται αυτό μετά την μεταφορά, όπως έγινε με την οδηγία για τις υπηρεσίες, αυτό που χρειαζόμαστε είναι η ορατότητα ε, η γνωστοποίηση για τις ενδιαφερόμενα μέλη, μέρη, για τις εταιρείες, τους εργοδότες, τους εργαζόμενους. Θα ήταν καλύτερα αν ε, στις συναντήσεις των clusters μπορούσαμε να μοιραστούμε την εμπειρία και τα προβλήματα ε, για αυτούς για τους οποίους εκπονείται ο νόμος ο νόμος ε, που ε, θεσπίζεται σε ευρωπαϊκό επίπεδο και μετά μεταφέρεται στην εθνική νομοθεσία. Αυτό θα διευκόλυνε ε, καλύτερη κατανόηση και καλύτερη κατάσταση στο μέλλον. Όσον αφορά την ερώτηση του κυρίου Σβάμπ, θεωρούμε την εμπειρία που αποκτήσαμε από την εργασία σε clusters με την Γερμανία ότι έτσι γνωριζόμαστε καλύτερα και μπορούμε να εξηγήσουμε ε, σε όλους την εταιρεία γιατί τα πράγματα και στους εταιρείες σας, στους εργαζόμενους, γιατί τα πράγματα έχουν ως έχουν. Αυτή η συνεργασία μεταξύ εθνικών δικήσεων είναι πάρα πολύ πολύτιμη διότι εμείς οι ειδικήσεις μετά πρέπει να επιλύσουμε τα προβλήματα των εταιριών και των ατόμων. Αυτή η εργασία σε clusters, κυρίως χωρών που έχουν μαζί ε, επιχειρήσεις και συνεργασίες και που είναι γειτονικέ χώρες, είναι πολύτιμη εμπειρία που αποφέρει καλά αποτελέσματα για το μέλλον. Euh, Είχα προβλέψει να αναφερθώ σε διάφορα σημεία. Θα έχω και την δεύτερη παρουσίαση, θα επανέλθω, κυρίως για το θέμα της διαφάνειας των εταίρων, ε, των ενδιαφερομένων μερών. Εδώ ήθελα ίσως να αναφερθώ σε αυτά που λέχθηκε για το τι συμβαίνει, θα συμβεί μετά σε 3, 4, 5 χρόνια για να κρατήσουμε τα όσα μάθαμε στην περίοδο αμοιβαίας αξιολόγησης. Θα σας πω ποια είναι η θέση της Γαλλίας ως προς το θέμα αυτό. Ήδη υπήρχαν πάρα πολλά έγγραφα εργασίας που εκπονήθηκαν και στις Ολομέλειες. Υπάρχει κάτι το γραπτό που παραμένει που είναι κάτι το σημαντικό και διαχρονικό. Εμείς, οι, οι Γάλλοι δηλαδή εμπειρογνώμονες, μπόρεσαν να συγχωνεύσουν τα όσα λέχθηκαν στις ομάδες. Η δίκηση η γαλλική λοιπόν έχει πλήρη γνώση. Και μετά, δεν ξέρω, αν άλλα κράτη-μέλη ακολούθησαν αυτόν τον ίδιο δρόμο, αποφασίσαμε ε, να έχουμε, αν θέλετε, πυρήνες κατά κάποιο τρόπο, που είναι πιο περιορισμένες ως προς την πλαισίωση από ό,τι είχαμε στις ομάδες ε, για την μεταφορά και την αμοιβαία αξιολόγηση. Αυτοί οι πυρήνες που, αν θέλετε, οι θεματοφύλακες ε, της οδηγίας. Αυτά για την αμοιβαία αξιολόγηση. Ε, κυρία Τραμπάχερ. Ευχαριστώ. Αντιλαμβάνομαι. Ευχαριστώ πολύ. Όσον αφορά ε, το τι θα γίνει στο μέλλον, τι θα κάνουμε στο μέλλον. Αυτό είναι ένα πάρα πολύ σημαντικό θέμα. Δεν πρέπει να ξεχάσουμε και δεν πρέπει να χάσουμε τη δουλειά που έχουμε κάνει στο παρελθόν. Όσον αφορά την ε, Σουηδία, ε, θεωρούμε ότι οι αποφάσεις για την οδηγία θα πρέπει να είναι αποφάσεις οι οποίες θα ληφθούν με τρόπο υπεύθυνο και που θα αφορούν ολόκληρη την οργάνωση γύρω από τα στην οδηγία προβλεπόμενα. Είναι σημαντικό το τι θα αποφασίσουμε να κάνουμε. Υπάρχουν νέα πράγματα τα οποία ενδεχομένως θα πρέπει να γίνουν και τα οποία θα σκεφτούμε σιγά σιγά στο μέλλον. Ε, ε, όπως έλεγε και η Γαλλίδα συνάδελφος ε, θα παραμείνει μια ε, λειτουργική ομάδα η οποία θα είναι η δικιά μας ευθύνη και θα πρέπει όλοι να κατανοήσουν και να βοηθήσουμε και εμείς να κατανοήσουν όλοι το περιεχόμενο της οδηγίας για τις υπηρεσίες. Το σημείο αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Είχαμε αποφασίσει στις, φάσεις, στις φάσεις αξιολόγησης είχαμε αποφασίσει λέω να δημιουργήσουμε μια ειδική ομάδα η οποία θα μπορούσε να συμμετάσχει στις διαπραγματεύσεις. Μια ε, ειδική ομάδα λέω ε, ε, ενδιαφερομένων stakeholders με εργαζόμενους, με business organizations, με προσώπους εργοδοτών και μάλιστα ε, θέλαμε οι επαφές μεταξύ τους να είναι τακτικές. Στη διάρκεια της προετοιμασίας ε, προσπαθήσαμε να καταλάβουμε ε, ποια ήταν τα κυριότερα μελήματα όλων των εμπλεκομένων φορέων για την εσωτερική αγορά και πιστεύουμε ότι οι ανταλλαγές αυτές είναι ένα πολύ σημαντικό input, μπορούν να μας διευκολύνουν τη δουλειά μας. Εμείς λοιπόν καλέσαμε τακτικά ε, τους εμπλεκόμενους φορείς στη διαδικασία αυτή. Δεν ξέρω ποια ήταν η δικιά τους άποψη, αλλά κατά την άποψή μας ε, αυτή η διαδικασία ανταλλαγής ε, με τους εμπλεκόμενους φορείς ήταν πάρα πολύ θετική. Όσον αφορά το κλάστερ μας, δουλέψαμε με την Εστονία, τη Λετωνία, τη Λιθουανία και την Φιλανδία. Δημοκρατίες Βαλτικής λοιπόν και Φιλανδία και Σουηδία. Ε, συναντηθήκαμε αρκετές φορές, μιλήσαμε για θέματα μεταφοράς ε, στο Εθνικό Δίκαιο. Αντιμετωπίσαμε τους τρόπους εφαρμογής ε, της οδηγίας, προσπαθήσαμε να καταλάβουμε τι κάνανε οι άλλες χώρες και είχαμε πολύ καλές ανταλλαγές οι οποίες ε, πάρα πολύ βοήθησαν την δουλειά μας. Όσον αφορά τα κλάστερ πρέπει να πω ότι δεν είχαμε προβλήματα και δεν έχω και κάποιε άλλε παρατηρήσει να κάνω. Well, Σας ευχαριστώ πολύ. Βρήκαμε νομίζω πάρα πολλές ενδιαφέρουσες πληροφορίες σε αυτό που μας είπατε. Είχαμε δύο στάδια ε, στο, ερωτηματολόγιο μας. Δεν έχω δώσει ακόμα το λόγο στην ε, εκπρόσωπο της Κομισιόν, γιατί θέλω να έχει τη δυνατότητα να κάνει μια αναθεώρηση του πρώτου τμήματος και να μας κάνει εισαγωγή του δευτέρου, που είναι η αξιολόγηση του κατά πόσον αυτή η αμοιβαία αξιολόγηση μπορεί να είναι ένα μέσο για την βελτίωση της λειτουργίας της ε, αγορά γενικά. και πώς μπορεί να εφαρμοστούν όλα αυτά εύκολα μπορούν όλα αυτά να εξεταστούν Η άποψη της ε, κυρίας Κεφάρτ ήταν πάρα πολύ σημαντική για την μνήμη των ε, οργάνων που ασχολήθηκαν με το θέμα αυτό. Και μετά θα πρέπει να δούμε κατά πόσον οι δημόσιες ε, διοικήσεις μπορούν να συνεργαστούν στο μέλλον για να μπορούν να εφαρμόσουν κάποια από τα στοιχεία αυτά πιο ευρέω. Έχουμε παραδείγματος χάρη την ε, ε η υπηρεσία ενημέρωση τη αγοράς, αγορά, την οποία θα συζητήσουμε κάτι... ε, αύριο, κατά σύμπτωση. Μπορείτε λοιπόν να κάπως να αναθεωρήσετε, να σχολιάσετε κυρία Μπρούμτερ Κόρετ αυτά που ακούσατε μέχρι στιγμής και να μας κάτι εμείς στο δεύτερο τμήμα. Να επανέλθουμε σε ερωτήσεις και τα θέματα που τέθηκαν για να απαντήσω στην κυρία Γκέμπερτ ε, για τι θα γίνει, τι θα συμβεί σε τρία χρόνια. Βεβαίως για την οδηγία για τις υπηρεσίες ελπίζουμε ε, για την δεκαετία που θα έρθει την επόμενη εβδομάδα θα ωφελούμαστε ακόμα ε, και από την γνώση και την ε, δικτύωση ε, της αμοιβαία αξιολόγησης και κάθε φορά που θα επανερχόμαστε με ορισμένες προτάσεις και συζητήσεις με κράτη-μέλη, αυτή η αμοιβαία κατανόηση ελπίζουμε ότι θα διευκολύνει τη συζήτηση διότι θα υπάρξει περισσότερη αμοιβαία κατανόηση, αμοιβαία εμπιστοσύνη αν θέλετε και θα μπορούμε να κάνουμε κάποια πρόοδο. Έχουμε ε, μεγάλο πρόγραμμα εργασίας ε, που μπορούμε να αγγείλουμε μετά την αμοιβαία αξιολόγηση που θα πρέπει να ακολουθήσουμε σύντομα με τα αποτελέσματα σχετικά ε, με την δυνατότητα να υπάρξει μια τέτοια διαδικασία πριν από την μεταφορά αυτό θα επιφέρει κάποια σύγχυση εάν κάνουμε αυτή την αμοιβαία αξιολόγηση κατά τη διάρκεια της μεταφοράς για πολλούς λόγους, ένας από τους οποίους είναι ότι η διαδικασία χρησιμοποιήθηκε για την αξιολόγηση του πώς τα κράτη-μέλη χρησιμοποίησαν την, το περιθώριο που είχαν για την οδηγία και όπως λέχθηκε από την εκπρόσωπο των Βρυξελών ε, πρέπει οι πολιτικές αποφάσεις να λαμβάνονται σε εθνικό επίπεδο επίσης. Είναι πάρα πολύ ε, δύσκολο λοιπόν αν δεν έχετε να συζητήσετε με τους άλλους, αν δεν έχετε αποφασίσει σε επίπεδο κοινοβουλίου ποια θα είναι η λύση όταν έχετε ένα μεγάλο περιθώριο ελιγμού είναι λοιπόν δύσκολο να προβλέψει, να προδικάσει κανείς αυτές τις συζητήσεις όταν τα μέρη δεν θα έχουν αρκετά βεβαιότητα για την πολιτική επιλογή και επιπλέον μπορεί να υπάρξει κίνδυνος να ξανανοίξουν διαπραγματεύσεις που έχουν λάβει χώρα σε επίπεδο Συμβουλίου για την υιοθέτηση της οδηγίας. Προσωπικά αυτό θα μπορούσε να ε, θέσει σε κίνδυνο την, ε, τον χρόνο της ε, μεταφοράς και τα αποτελέσματα από τα κράτη-μέλη σχετικά με την μεταφορά. Δεν πιστεύουμε λοιπόν ότι ως γενική αρχή θα πρέπει να υπάρχει με τέτοια διαδικασία πριν. Τώρα, σχετικά με την ερώτηση της κυρίας Χάνσλι αν θα χρησιμοποιήσει η Κομισιόν τα αποτελέσματα της αμοιβαίας αξιολόγησης, ούτω ώστε να ε, ενισχύσει την ε, οδηγία για τις υπηρεσίες. Υπήρξε μια κατανόηση εκ μέρους μας και δέσμευση ότι δεν ήταν αυτός ο στόχος και δεν θα πρέπει ούτε καν ε, να είναι η συνέπεια. Γι' αυτό η Κομισιόν δεν το έπραξε και για τον απλό λόγο ότι η Κομισιόν είχε όλα τα μέσα για να εξετάσει τα εθνικά κείμενα, κυρίως και σε όλες τις γλώσσες και αν νομίζαμε ότι ε, υπήρχαν ε, παραβάσεις, αυτό που θα μπορούσε να γίνει ανεξάρτητα από την διαδικασία αμοιβαία αξιολόγησης. αν πιστεύει η Κομισιόν ότι ένας περιορισμός δεν είναι πλέον δικαιολογημένος, τότε αναλαμβάνει ευθύνη να ανοίξει την διαδικασία επί παραβάση. Ακούγοντας την Région Bruxelles Capital, επιμένουμε περισσότερο πάνω σε αυτό, διότι φαίνεται ότι η παρουσία μας θα μπορούσε να δημιουργήσει δυσκολία για την ανταλλαγή και βεβαίως η Κομισιόν δεν χρησιμοποίησε τα αποτελέσματα της αμοιβαία αξιολόγησης ως μέσο ελέγχου ε, των μέτρων μεταφοράς. Και τέλος, ήταν ενδιαφερόμενα μέρη και η διαφάνεια, αυτό που είπε ο εμπειρογνώμων ήταν ενδιαφέρον με την έννοια ότι πιθανόν ο καλύτερος τρόπος να οργανώσει κανείς την αμοιβαία αξιολόγηση και την έλεγχο. Αυτό μπορεί να γίνει και σε εθνικό επίπεδο. Τα ενδιαφερόμενα μέρη από τα διάφορα κράτη-μέλη, αν πολλαπλασιάσουμε με τον αριθμό των ενδιαφερομένων μερών από κάθε κράτος μέλος θα είναι πάρα πολλά τα άτομα και δεν βλέπουμε πώς το σύστημα θα μπορούσε να λειτουργήσει. Κάναμε ό,τι μπορούσαμε σε επίπεδο ευρωπαϊκό. Υπήρξαν μόνο ευρωπαϊκές ομοσπονδίες και εκπρόσωποι σε ευρωπαϊκό επίπεδο που συμμετείχαν, αλλά πιστεύουμε ότι τα κράτη-μέλη κάνουν το ίδιο σε εθνικό επίπεδο κατά τη διάρκεια της ίδιας της διαδικασίας και αυτός ο συνδυασμός θα μπορούσε βεβαίως να βελτιώσει ε, την ε, διαφάνεια για τα ενδιαφερόμενα μέρη. Αυτό με οδηγεί τώρα ε, στο δεύτερο μέρος της ακρόασης που σχετίζεται με την ε, χρησιμοποίηση της αμοιβαίας αξιολόγησης ως εργαλείο, θα έλεγα, διότι δεν μπόρεσα να το πω στην πρώτη παρέμβαση, ότι από την άποψη της Επιτροπής αυτή η αμοιβαία αξιολόγηση ήταν για μας μια χρήσιμη άσκηση και ότι άξιζε την προσπάθεια. Δεν θα είχαμε ε, τέτοια γνώση, βαθιά γνώση ε, ε, για το πώς λειτουργεί η οδηγία χωρίς αυτή τη διαδικασία. Χωρίς. Σαφώς ε, πρόκειται για κάτι το θετικό, κάτι που έχουμε στο ενεργητικό μας, αλλά πάντοτε υπήρξαμε σαφείς για το ότι η αμοιβαία αξιολόγηση δεν πρέπει να χρησιμοποιείται με συστηματικό τρόπο ούτε ως μόνο μέσο για την αξιολόγηση της υλοποίησης της οδηγίας. Και νομίζω ότι το αναφέραμε αυτό και στην ανακοίνωση ε, και αλλού, όπου ε, δεν ε, αποφαινόμαστε ότι πρόκειται για μία πρότυπη κανονική διαδικασία. Ξετάζοντας την έκθεση των εμπειρογνωμόνων, βλέπουμε ότι τα κριτήρια που προτάθηκαν στην έκθεση ε, έχουν σημασία. Πρώτα απ' όλα θα έπρεπε να τα χρησιμοποιήσουμε για τους οδηγίες, όχι για τους κανονισμούς ε, και για οδηγίες πλαίσιο. Η οδηγία για τις υπηρεσίες είναι ένα καλό παράδειγμα ε, του πεδίου εφαρμογής που είναι το κατάλληλο. Μπορούμε να τη χρησιμοποιήσουμε όταν δίνεται κάποια ελευθερία στα κράτη-μέλη, κάποιο περιθώριο και ήταν εδώ η περίπτωση για την οδηγία για τις υπηρεσίες και όταν αυτό γίνεται ε, για στρατηγικές ε, διατάξεις σε τομέα που είναι σημαντικός για την εσωτερική αγορά και πάλι δεν πιστεύουμε ότι ε, πρέπει σε άλλη φάση να χρησιμοποιείται αυτή η διαδικασία. Αυτό πρέπει να είναι μια διαφορετική άσκηση από ότι ο έλεγχος της μεταφοράς από τα κράτη-μέλη. Είμαστε καλά εξοπλισμένοι για να ελέγξουμε τη μεταφορά στην εθνική νομοθεσία. Έχουμε ε, συνεργασίες διάφορες της Κομισιόν με τα κρατημέλη και για μας η αμοιβαία ε, αξιολόγηση μας μαθαίνει πολλά πράγματα, πρέπει να περιορίζεται ειδικά σε ορισμένα ε, κείμενα Ε, πρέπει σε άλλες περιπτώσεις να υπάρχει διερευνητική εργασία. Βεβαίως πρέπει να λαμβάνουμε υπόψη το κόστος των πόρων τόσο για τα κράτη-μέλη όσο και για την Κομισιόν. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ πάρα πολύ σαφή όλα αυτά. <clears throat> Αυτό που θα κάνουμε θα πάμε πάλι πίσω στους εμπειρογνώμονες μας ή έχουν κάποια στοιχεία να προσθέσουν να μας πούνε τι πιστεύουν για την εφαρμογή του συστήματος σε άλλους τομείς. είναι πολύ προκλητική η ερώτηση, ε, αλλά επειδή έχετε πείρα στον τομέα των βεσιών, θα μπορούσατε να μας πείτε τι φαντάζεστε ε, για την εφαρμογή σε άλλους τομείς. Ο κύριος Λεπλά, ε, αλλά να αρχίσουμε με την κυρία Μασάρ να απαντήσει πρώτα εκείνη και μετά θα πάμε ένα προς ένα. Η κυρία Μασάρ να απαντήσει. Είχα υποσχεθεί να απαντήσω και σε κάποιες ερωτήσεις που υποβλήθησαν. Ξέρω πώς θα το κάνω τώρα. Κοιτάξτε, είναι αυτές οι συζητήσεις μεταξύ των ε, κρατών ε, με ελευθερία λόγου, με διαφάνεια. Τονίζω αυτό το σημείο ιδιαίτερα και γι' αυτό υπήρχε η αναγκαιότητα ε, του απορρίτου κατά κάποιον τρόπο των εργασιών. <clears throat> Αυτή, αυτό το απόρριτο ήταν απαραίτητο για να υπάρχει η δυνατότητα ελευθέρων και ηλεκτρονών συναλλαγών. Ελέγχθη το θετικό είναι ότι έτσι μπορεί να γνωρίσει κανένας ε, την ομοθεσία των άλλων κρατών, ότι μπορεί να ωφεληθεί από εναλλακτικά μέσα, από ε, εναλλακτικά πρότυπα που χρησιμοποιούνται αλλού, να γνωρίσει καλές πρακτικές. Μετά την μεταφορά της νομοθεσίας είναι σημαντικό. Αυτά είναι όλα θετικά. Τώρα όσον αφορά τα αρνητικά στοιχεία της διαδικασίας αμοιβαίας ε, αξιολόγηση είναι το διοικητικό τμήμα γιατί κινητοποιεί πολύ προσωπικό. Στη Γαλλία διατηρήσαμε την ίδια ομάδα εκείνη που είχαμε για τη μεταφορά της οδηγίας και επίσης το ίδιο δίκτυο αν θέλετε, ε, συνομιλητών μας στα διάφορα υπουργεία, όπως υπήρχαν προηγουμένως. Αυτό κοστίζει βέβαια. αλλά πρέπει να το λάβουμε υπόψη στις επόμενες οδηγίες. Όσον αφορά τις βελτιώσεις. Η αμοιβαία αξιολόγηση στα πλαίσια οδηγίας της υπηρεσίας ήταν μια σύγκριση και θα ήταν πιστεύω ενδιαφέρον να συμπεριληφθούν συγκεκριμένες περιπτώσεις. Κάποια σενάρια. Όπως θα γίνει τώρα αυτό με την εξέταση της απόδοσης που προαναγγείλει η Κομισιόν. Αλλά αυτό είναι κάτι που θα μπορούσε να γίνει εκ μιας αρχής στην ίδια τη διαδικασία. Όσον αφορά τώρα το θέμα, κατά πόσον η αμοιβή αξιολόγηση θα πρέπει να γίνει πριν ή μετά τη μεταφορά. τέλο πάντων κατά τη διάρκεια τη μεταφορά ή μετά τη μεταφορά. Εγώ δεν έχω εκεί αποφασισμένη θέση. Υπάρχουν επιχειρήματα υπέρ και κατά και από τις δύο πλευρές. Θα μπορούσα όμως να φανταστώ ότι η κατεύθυνση μεταφοράς δεν έχουμε ακριβή και πλήρη εικόνα της νομοθεσίας που θα ενταχθεί ε, στα πλαίσια αυτής της οδηγίας. Υπάρχουν ακόμα εσωτερικά ερωτηματικά, υπάρχουν πολιτικές αποφάσεις που πρέπει να ληφθούν στο εθνικό επίπεδο. Και αυτό είπε και η κυρία Ζώ. Και όλα αυτά δεν μπορούμε να τα αξιολογήσουμε εκ των προτέρων. Τώρα, πού θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί η διαδικασία αυτή της αμοιβαίας αξιολόγησης, εδώ συμφωνώ με την Κομισιόν και με τους κυρίους Μπερζέ και Λεπλά, ότι δεν μπορεί να έχουμε συστηματική προσέγγιση. για τους άλλους τομείς. Δηλαδή καμιά φορά υπάρχουν οδηγίες με πολύ καθορισμένο πεδίο εφαρμογής. Εκεί δεν υπάρχει τόσο πολύ ενδιαφέρον για κάτι τέτοιο. Θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί για οδηγίες που έχουν ευρύ πεδίο εφαρμογής, όπου υπάρχουν δηλαδή για τα κράτη-μέλη ε, περιθώρια εκτίμησης και αξιολόγησης. Κατά γνώμη μου μόνο σε αυτό το πλαίσιο μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε αυτό το μέσο. Τελειώνω, Πρόεδρε. Όσον αφορά το θέμα των πινάκων προσέγγισης, νομίζω ότι το μεν δεν αποκλεί το δε, δηλαδή την αμοιβή αξιολόγηση. Αυτά τα, αυτοί οι πίνακες σύγκλησης στη Γαλλία κάναμε μια ε, ανατομέα αξιολόγηση κατά περίπτωση και να βρούμε εκεί ένα πίνακα σύγκληση θα ήταν πάρα πολύ ε, δύσκολο και δεν θα ήταν και καθόλου ευανάγνωστο τελικά. Ευχαριστώ. Πρώτα σας ευχαριστώ πολύ για σαφείς παρατηρήσεις που κάνατε και μας υπενθυμίστε και τα τέξ απόδοση, τα απόδοσης. Είναι πολύ ενδιαφέρον. Η κυρία Χάντλεκ θα τα σημειώσει. Η κυρία Βουίλ ε, θα το κάνω αυτό, θα σας πω Βουίλ μόνο. Ευχαριστώ. Θα ήθελα στα σύντομα να αναφερθώ σε αυτό που είπε η κυρία Παμέλα Μπράμτερ όσον αφορά την χρήση της ε, αμοιβαίας αξιολόγησης ή το τι θα σημαίνει αν δεν την είχαμε χρησιμοποιήσει για τη μεταφορά της οδηγίας. Έχουμε παραδείγματα και αναφέρεται στην έκθεση ότι υπάρχουν κάποιες χώρες, παραδείγματος χώρες στις σκανδιναβικές χώρες, που εργάζονται κατά διάρκεια της μεταφοράς στις ε, εναλλακτικέ ε, της μεταφοράς που θα θέλανε να χρησιμοποιήσουν στις διάφορες χώρες. Εάν είχαμε λοιπόν την ευκαιρία να συζητήσουμε τις διάφορες επιλογές για τη μεταφορά στα clusters, θα ήταν για αμοιβαίο, προς αμοιβαίο όφελος. Τώρα κατά πόσο μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε την αμοιβαία αξιολόγηση. Αυτό εξαρτάται νομίζω από τον τρόπο με τον οποίο αξιολογούμε αν θέλετε την αμοιβαία αξιολόγηση. Δηλαδή, εάν θεωρήσουμε ότι μπορούμε να τη χρησιμοποιήσουμε κατά τη διάρκεια της μεταφοράς με τη συμμετοχή των άμεσα ενδιαφερομένων πιστεύω ότι υπάρχουν πολλοί τομεί πολιτική στην εσωτερική αγορά που θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί κάτι τέτοιο. Εάν από την άλλη μεριά το σφαιρικό αποτέλεσμα της συζήτηση είναι ότι η αμοιβαία αξιολόγηση με, πρέπει να γίνει μετά τη μεταφορά για μια διαδικασία ε, εξερεύνησης των δεδομένων θα πρέπει να χρησιμοποιείται τότε άλλα περίπτωση. Ανάλογα με το σφαιρικό χαρακτήρα της οδηγίας, δηλαδή κατά πόσο είναι μια μεγάλη οριζόντια πολυπολιτική οδηγία, όπως αυτή η οδηγία για τις υπηρεσίες, τότε θεωρώ ότι η διαδικασία του να αποκτήσουμε καλύτερες γνώσεις της προσέγγισης των κρατών μελών είναι πολύ χρήσιμη. Αλλά το να χρησιμοποιηθεί η αμοιβαία αξιολόγηση για πιο απλή και άμεση οδηγία δεν νομίζω ότι είναι πολύ χρήσιμο. Ευχαριστώ πολύ. Νομίζω ότι οι συνάδελφοί μου τα είπαν όλα, αλλά και από τις προηγούμενες παρεμβάσεις μου θα καταλάβατε ότι τη στιγμή της ε, αμοιβαίας αξιολόγησης είχαμε έτσι κάποια ερωτήματα. Γιατί όταν σκεφτόμαστε ποιοι είναι οι στόχοι της διαδικασίας που θέλουν να οδηγήσουν σε, δημιουργία μιας ειδική δυναμικής, κατανοούμε ότι δεν πρόκειται μονάχα για ένα τεχνικό εργαλείο, είναι και πολιτικό εργαλείο. Και εγώ το βλέπω καθαρά ε, στην περιφέρεια για την οποία εργάζομαι, μία από τις άμεσες ε, επιπτώσεις ε, είναι η σταθεροποίηση, η σταθερότητα μιας ε, ομάδας η οποία θα δουλέψει για αυτό το σκοπό και μπορεί να έχει μια, έναν ειδικό αντίκτυπο, σημαντικό μάλιστα. Μια και όντως έχουμε επενδύσει ε, σε κόστος, σε ανθρώπινο ε, υλικό και επομένως σε ανθρώπινους πόρους και επομένως θα συνεχίσουμε να επενδύουμε. Τώρα, ε, σε σχέση με άλλους τομείς και την, το ενδεχόμενο να διευρυνθεί η διαδικασία και σε άλλους τομείς δεν νομίζω. Δεν έχω όμως προσωπική άποψη, απλώς πιστεύω ότι είναι μια διαδικασία η οποία θα πρέπει να συνδέεται με συγκεκριμένες πολιτικές δράσεις, ας πούμε, όπως πράξη για την ενιαία αγορά. Αυτά ήθελα να πω. Ευχαριστώ. Ε, Κυρία Γκέμπχαρτ. Comme nous l'indiquons dans notre rapport, il est à notre sens prématuré de pouvoir... Ο, συγγνώμη, ο κύριος Λεπά. κατανοήσαμε ε, συζητώντας για τη γενίκευση της ε, διαδικασίας ε, ότι μια κύρια επίπτωση ήταν η καλύτερη κατανόηση της χρήσης αυτού του εργαλείου για καλύτερη κατανόηση της, των, των μονάδων, των υπηρεσιών και βεβαίως της ίδιας της ενιαίας αγοράς. Αυτά. Δύο λόγια. Δύο λόγια λοιπόν για τη διαδικασία. Ε, βεβαίως μπορούμε να πάρουμε το τυπικό σκέλος, να πούμε ότι στις οδηγίες πλαίσιο υπήρχαν οι στρατηγικές αναλύσεις, αλλά μπορώ να πω δύο λόγια. Πρώτα απ' όλα η διαδικασία είναι εξαιρετικά χρήσιμη για όλα τα στοιχεία τα οποία παρουσιάζουν εξελικτικό χαρακτήρα και νομίζουμε ότι ακριβώς ε, η ευρωπαϊκή πολιτική βασίζεται στην εξελικτική διαδικασία και είναι κατά κάποιο τρόπο ο μύτος της Αριάδνης που θα μας ακολουθήσει σε όλες τις ε, περιπτώσεις. Ε, για να συμμετάσχουν τα κράτη σε αυτή τη διαδικασία. Έτσι έχουν επιλεχθεί και τα ερωτήματα μέσα στα πλαίσια της οδηγίας για τις υπηρεσίες ότι δεν υπήρχε συνένεση για τις λύσεις τελικά. Υπήρχαν προβλήματα σχετικά. Το δεύτερο που θα μπορούσε να είναι κριτήριο ουσιαστικό, όχι τυπικό, είναι το θέμα της δυνατότητα συνεργασία. Και εγώ θα αναφερθώ σε ένα άλλο τομέα που δεν σχετίζεται με την Επιτροπή αυτή, αλλά που αναφέρθηκε προηγουμένω. Ε, ελευθερία, ασφάλεια, δικαιοσύνη. Σε αυτές τις περιπτώσεις ε, η συνεργασία ειδικά μεταξύ δικαστών ε, εθνικών αρχών που ενέχονται ότι στον χώρο ελευθερίας και δικαιοσύνης ε, είναι κάτι πάρα πολύ σημαντικό γιατί δεν γνωριζόμαστε και άρα δεν έχουμε εμπιστοσύνη. Η εμπιστοσύνη όμως είναι η λέξη κλειδί ακριβώς ε, όσον αφορά την αμοιβαία αναγνώριση και την αμοιβαία ανεξιολόγηση και επομένως ε, ορίστε ένα θετικό στοιχείο το οποίο είναι ε, καλό για την οικοδόμηση της ενίας αγοράς. Επανέρχομαι λοιπόν σε αυτό που έλεγα και προηγουμένως, δηλαδή ότι ενδεχομένως θα πρέπει να λειτουργήσουμε ε, ε, ευνώντας ακόμα περισσότερο όλα αυτά τα εργαλεία τα οποία είναι εργαλεία συνεργασίας και που θα δώσουν την δυνατότητα να συνεννοηθούν καλύτερα, να συναντηθούν και να γνωριστούν οι εκπρόσωποι των διαφόρων υπηρεσιών έτσι ώστε να χτιστεί η απαραίτητη εμπιστοσύνη και έτσι να ανοιχτεί ένας καινούργιος δρόμος για το μέλλον της αμοιβαίας αξιολόγησης. Ευχαριστώ. παρακαλώ. Τελευταία. Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε. Θα ήθελα να ξεκινήσω με την ε, ερώτηση που κάνατε, δηλαδή εάν αυτή η αμοιβαία αξιολόγηση μπορεί να χρησιμοποιηθεί και σε άλλους τομείς. Η απάντησή μου είναι πάρα πολύ απλή. Εξαρτάται. Εξαρτάται από το πεδίο εφαρμογής, εξαρτάται από την, ε, από την δομή, εξαρτάται από το ποιο είδος, ποια μορφή πολιτικής στήριξης ε, έχουμε. Ε, ε, εξαρτάται. Γενικώ πρέπει να παρακολουθήσουμε από κοντά την κάθε περίπτωση για να απαντήσουμε. Βεβαίως υπάρχει η δυνατότητα να δούμε εάν μπορούμε και να επαληθεύσουμε αν αυτή η αμοιβαία αξιολόγηση πέραν της οδηγίας για τις υπηρεσίες μπορεί να χρησιμοποιηθεί και αλλού. Γιατί θεωρώ ότι ήταν θετική η εμπειρία της οδηγίας για τις υπηρεσίες, μα το είπαν ήδη προναλύσαντες είναι σημαντικό να γίνεται λόγος ε, για την αναλογικότητα. Η οδηγία για τις υπηρεσίες είναι μια περίπλοκη οδηγία. Είναι πάρα πολύ σημαντικό λοιπόν, ε, ήταν σημαντικό που είχαμε την δυνατότητα να συζητήσουμε, να συζητήσουμε στα πλαίσια της αξιολόγησης το θέμα της αναλογικότητας. και επίσης ε, να ασχοληθούμε με κάποια συγκεκριμένα κριτήρια τα οποία μας επευλήθησαν αλλά μας οδήγησαν παρόλα αυτά σε κάποια πολύ θετικά συμπεράσματα. Νομίζω ότι ξεκινώντας ε, να δουλεύουμε σε ομάδες κατανοούμε καλύτερα την αρχή της αναλογικότητας. Δημιουργήθηκαν λοιπόν ομάδες στα πλαίσια ε, της ε, διαδικασίας αξιολόγησης ε, στην οδηγία για τις υπηρεσίες. Δημιουργήθηκαν λέω ομάδες οι οποίες έδωσαν μια νέα όθηση στο θέμα της εμπιστοσύνης και της αμοιβαίας αξιολόγησης. Ξέρετε, δεν ήταν πάντα ε, ε, πολύ ευχάριστο ή εύκολο το να ασχολούμαστε με τα επιμέρους ε, προβλεπόμενα από την οδηγία για τις υπηρεσίες. Οι ανταλλαγές όμως ήταν πάρα πολύ σημαντικές. Πολλοί είχαν το θάρρος να απευθύνουν ερωτήσεις και πολλές φορές ερωτήσεις οι οποίες ήταν δύσκολες, μας έφεραν σε δύσκολη θέση και επίσης πολλές φορές και η ίδια η Επιτροπή πρόωθησε κάποιες συζητήσεις στα πλαίσια της Ολομέλειας. Χωρίς τις συζητήσεις αυτές δεν θα μπορούσαμε να είχαμε αυτά τα εξαιρετικά αποτελέσματα. Όσον αφορά την άλλη ερώτηση, δηλαδή αν θεωρούμε ότι αυτή η διαδικασία ε, θα έπρεπε να έχει λάβει χώρα πριν. Όπως είπε και η Γαλλίδα συνάδελφος, πιστεύω ότι εάν δεν υπάρχει τίποτα στο τραπέζι, ε, δεν μπορούμε να ξεκινήσουμε Πρέπει να ξέρουμε, πρέπει να έχουμε κάποιες αρχές που να μας οδηγούν. Πάντως μας οδήγησε σε καλύτερη συνεργασία ε, με, τουλάχιστον για το δικό μας κλάστερ, με τους γείτονές μας, με τις χώρες της Βαλτικής, της Δημοκρατίας της Βαλτικής και αυτό ήταν πάρα πολύ θετικό. Νομίζω ότι θα ήταν δύσκολο να κάνουμε μια τέτοια διαδικασία μετά την έγκριση της οδηγίας. Ευχαριστώ. Να σας ευχαριστήσω όλους που μοιραστήκατε μαζί μας τις απόψεις σας. Έχουμε ακόμα λίγο χρόνο. Θα πω στην κυρία Γκέπχαρτ αν θέλει να εξάγει κάποια πρώτα συμπεράσματα ε, και μετά η κυρία και ενδεχομένως ε, να κάνει τις δικές της τελικές σκέψεις. Η κυρία Γκέμπχαρτ πρώτα. Ευχαριστώ. Και θέλω να σας ευχαριστήσω την καρδιότητα και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και τους εμπεργνώμενους που ήρθαν εδώ, που ήταν πάρα πολύ ικανοί και μας έδωσαν τόσες πολλές πληροφορίες και που αναφέρθηκαν συγκεκριμένα στα ερωτήματα ε, που είχαμε υποβάλει και μας απάντησαν σε αυτά. Δεν συμβαίνει σε κάθε ακρόαση αυτό και γι' αυτό, αυτό φαίνεται ότι είναι πάρα πολύ θετικό. με έκανε και εμένα να ξανασκεφτώ κατά πόσο θα πρέπει να είμαι τόσο πια σκεπτική εναντί αυτού του συστήματος της ε, αμοιβίας αξιολόγησης. Ε, οπωσδήποτε μπορούμε να το γενικοποιήσουμε γιατί το κόστος είναι πάρα πολύ ψηλό, οι απαιτήσει είναι πάρα πολύ ψηλές και πρέπει να χρησιμοποιείται με μέτρο στις περιπτώσεις δηλαδή που μπορεί να χρησιμοποιηθεί ε, προς όφελος ε, της διαδικασίας μεταφοράς της νομοθεσίας. Έχω μία μικρή, μικρή ερώτηση, ε, γιατί νομίζω ότι ένα από τα ερωτήματα της κυρίας Άσλικ δεν απαντήθηκε ακόμα και θα ήθελα να προσθέσω κάτι. Ίσως η κυρία Βίλι ή η κυρία Στραντπακ ε, μπορεί να απαντήσουν για τα κλάστερ. Ε, φαίνεται ότι είναι γραφικής μορφής είχατε τη δυνατότητα εσείς να συναποφασίσετε τι μορφή θα είχαν, τι σύνθεση θα είχαν. Θα ήταν επίσης ενδιαφέρον στα κλάθη αυτά να υπάρχουν και χώρες πιο απομακρυσμένες για να υπάρχει και ένα πιο ευρύ φάσμα ε, πολιτισμικό νοοτροπίας. Σουηδία και Ελλάδα, Φερρυπίν. Θα ήταν ένας συνδυασμός ήσασταν ικανοποιημένοι τελικά με τη διαδικασία αυτών των κλάστερ. Well, I mean, we could, I think we have just time. Η ε, κυρία Μπρόντον ήταν επικεφαλής της όλης διαδικασίας για τα κλάστερς. Ίσως θα πρέπει να ρωτήσουμε την Κομισιόν πώς διαμορφώθηκαν αυτά τα κλάστερς. Μήπως να απαντήσετε εν συντομία προτού κλείσουμε. λάβαμε την απόφαση σχετικά με τα κράτη-μέλη για τα clusters, αλλά το κάναμε αυτό με διαφορετικά κριτήρια, το επίπεδο των εμπορικών σχέσεων ανάμεσα στα κράτη, τη γλώσσα. Η γλώσσα ήταν επίσης ένα κριτήριο. Με βάση τα κριτήρια αυτά, Ε, εντάχθηκαν ε, σε κλάστερ και συμμετείχαν σε αυτά, σε αυτές τις συστάδες χωρών. Δεν ξέρω αν όλοι ήταν ευχαριστημένοι την ε, πρώτη στιγμή όταν έλαβαν τον κατάλογο, αλλά νομίζω ότι τελικά λειτουργήσε καλά το σύστημα και ήταν καλές οι ανταλλαγές με τα άλλα κράτη-μέλη του κλάστερ. Ίσως υπάρχουν άλλα κριτήρια που μπορεί να επιλεγούν για αυτή τη διαδικασία, αλλά όταν συζητήσαμε για μια αναμόρφωση των κλάστερς κατά τη διάρκεια της διαδικασίας, νομίζω, νομίσαμε και, το, και επικρότησαν και οι, ε, οι εμπειρογνώμονες ότι θα, το σύστημα θα γινόταν πολύ πιο περίπλοκο, καλύτερα να υπάρχει κάποια ευηλιξία στα clusters. Ίσως θα μπορούσαν ε, τα ίδια να αποφασίσουν, αυτό μπορεί να ήταν ε, κάποια ε, λύση. Αλλά κάποιος πρέπει να αποφασίσει τελικά για ένα τέτοιο θέμα. Γιατί ίσως όλα τα κρατημέλη θα ήθελαν να είναι στο ίδιο κλάστερ ε, με ορισμένους αφήνοντας μερικούς απομονωμένους μόνους τους. Ευχαριστώ πολύ. Νομίζω ότι η συγκήτριά μας θα συζητήσει μαζί σας. Μερικά λόγια για να κλείστε Πού πάμε από εδώ για να κλείσουμε τη συνεδρίαση. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Ευχαριστώ όλους τους εμπειρογνώμονες. Πιστεύω ότι ήταν μια πολύ καρποφόρα συνεδρίαση, επικοδομητική, μάθαμε πολλά ενδιαφέροντα πράγματα, λάβαμε πολλές πληροφορίες και χάρη στους συναδέλφους έλαβα όλες τις απαντήσεις στις ερωτήσεις μου. Είχαν ε, απάντηση για όλες τις ερωτήσεις. Βεβαίως αυτές οι πληροφορίες θα συμβάλλουν στην εχνομοδότησή μου, η οποία θα είναι πληρέστερη. Και κάτι κάποιο τρόπο θα είναι ευρύτερη. Αφού άκουσα τις απόψεις σας, θα μπορούσα να πω ότι αυτή η διαδικασία αμοιβαία αξιολόγησης παρά την αρνητική στάση απέναντί της στην αρχή, σχετικά με την οδηγία για τις υπηρεσίες, νομίζω ότι τελικά ήταν μια πολύ θετική εμπειρία για τα ίδια τα, ίδια τα κράτη-μέλη. Και εγώ πιστεύω ότι σε μεγάλο βαθμό συνέβαλε σε καλύτερη κατανόηση, θα έλεγα αμοιβαία κατανόηση ανάμεσα στα διάφορα κράτη-μέλη ε, για, ε, σχετικά με ορισμένα στοιχεία ε, που λείπουν από την διαδικασία υλοποίησης. Σας ευχαριστώ για την προσοχή σας και θα κλείσουμε αυτήν την δημόσια κρόαση. Θέλουμε να εκφράσουμε την ευγνωμοσύνη μας ε, για την αγαστή συνεργασία που είχαμε κατά τη διάρκεια αυτής της ακρόασης. Και πρωτού κλείσουμε τη συνεδρίαση θα ήθελα να σας κοινοποιήσω ότι ε, το πρόγραμμα είναι μέχρι τον, την 21η Ιουνίου θα έχει μεταφραστεί η εισήγηση και μετά στις 12 Ιουλίου θα εξεταστεί στο ε, σχέδιο 18 Ιουλίου για τις τροπολογίες. 30 Αυγούστου θα εξετάσουμε τις τροπολογίες ε, και στις 19 Σεπτεμβρίου θα ψηφιστεί και επίσης προγραμματίζουμε ε, ψηφοφορία στην Ολομέλεια του Οκτωβρίου στο Στρασβούργο της Γαλλίας. Αυτό είναι το πρόγραμμα, το χρονοδιάγραμμα που θα ακολουθήσουμε. Um, um, Ευχαριστώ όλους τους εμπειρογνώμονες. Ε, Βεβαίω θα εξετάσουμε λεπτομερό την μελέτη ο κύριος Μπεζιέ, ο κύριος Λεπλά. Τους ευχαριστούμε. Ελπίζω ότι ε, έχουμε αντίγραφα επίσης ε, για τους εμπειρογνώμονες αλλά ε, μπορείτε να συνεχίσετε να εργάζεστε πάνω σε αυτό το σημείο. Αν θέλετε να μας στείλετε παρατηρήσεις, είναι ευπρόσδεκτες. Θα ήθελα να έχουμε αυτό το, την εγκύκλιο για το δίκτυο που έχουμε για την ενιαία αγορά. Μπορείτε βεβαίως να συμβουλευτείτε το έγγραφο αυτό ε, στο διαδίκτυο, αλλά μπορείτε να λάβετε ε, και την, ένα αντίγραφο ως φίλοι του δικτύου. Ενθαρρύνουμε ε, τα μέλη των ομάδων αμοιβαίας αξιολόγησης επίσης ε, να ενδιαφερθούν για το δίκτυο αυτό. Ε, περιμένουμε την εισήγηση της κυρίας Χάνσλικ και η τελευταία μου παρατήρηση είναι ότι μερικά από τα σημεία που θίξαμε σχετικά με την ύλιοποίηση της οδηγίας για τις υπηρεσίες είναι κάτι που μπορεί να αποτελέσει μια μελλοντική εργασία και θα δούμε πόσο καλά γίνεται η εργασία, η συνεργασία και ποιες είναι οι δυνατότητες. Όλα αυτά τα πράγματα μας απασχολούν λόγω του σημαντικού όγκου εργασίας που, που κάνατε, χρειαζόμαστε αυτά τα αποτελέσματα και είπατε ότι με την εισήγηση θα έχουμε νέες δυνατότητες για τις αγορές την προώθηση των υπηρεσιών. Ευχαριστώ πολύ. Απλώς στα μέλη της Επιτροπής θέλω να πω ότι στις 9 η ώρα αύριο ξανασυνεδριάζουμε. Έχουμε ένα φορτωμένο πρόγραμμα αύριο, επίδειξη ε, για το σύστημα πληροφοριών ε, για την ε, εσωτερική αγορά. Ο Επίτροπος Τζον Ντάλι θα έρθει στις 9.30 για να μας μιλήσει για το μελλοντικό του πρόγραμμα. Θα έχουμε και μια άλλη ε, στις 10.30 μια μελέτη για την ουδετερότητα και μετά θα έχουμε την ψηφιακή ατζέντα. Θα έχουμε λοιπόν μια ενδιαφέρουσα συνεδρίαση. Ελπίζω να έρθετε πολύ πληθείς αύριο. Σας εύχομαι καλό βράδυ.